Να ξεκινήσουμε αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμοι, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, χαιρόμαστε που βρίσκεστε και πάλι μαζί μα. Ελπίζομαι να περάσατε καλά στι διακοπές, ε, να ξεκουραστήκατε και να φορτώσατε μπαταρίε για τι επόμενε εβδομάδε, τις ε, επόμενου μήνε, Από ό,τι βλέπω όλοι είσαστε σε εξαιρετική φόρμα και εγώ μια χαρά είμαι, ευτυχώ, λέει ο πρόεδρο. Και έτσι λοιπόν, να συγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσει. Τα πρακτικά τη 11η και 12η Ιουλίου 2016 επίση εγκρίνονται. Σε περίπτωση τουλάχιστον που δεν έχετε κάποια αντίρρηση. Ανακοινώσει του Πρόεδρου. Δεν έχουμε. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν με τι ε, ψηφοφορίε. Ε, Γενικό προπολογισμό του 2017. Η Ισαμπέλα Ντεμόντα είναι η συγγήτρια. Αλλά α κάνουμε και μια δοκιμαστική ψηφοφορία ηλεκτρονικά, να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Έναρξη ψηφοφορία παρακαλώ. Λαμβάνω γνώση, λέει ο πρόεδρο, δεν ξέρουμε ακριβώ τι, γιατί τα σχόλια ήταν εκτό μικροφώνου. Το έχουμε συνηθίσει. Θα τα βρούμε. Δεν λειτουργεί η συσκευή σα, συνάδελφε.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 5-9-2-8. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5-9-0-9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5-9-27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ζητείτε ηλεκτρονικός έλεγχος για την 5927. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. 17 υπέρ, 22 κατά. Καμία αποχή απορρίπτεται. Δεν θα λέω το 59, θα λέω μόνο τα δύο τελευταία ψήφια. 14 λοιπόν, υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται, μου φαίνεται, αλλά θα το ελέγξουμε. Έναρξη. Πέρας. 19 υπέρ, 22 κατά, απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. Για την 26, παρακαλώ, έναρξη. Πέρες. 27 υπέρ, 13 κατά. Σαφές. Ευχαριστώ αλλά το αποτέλεσμα ήταν, ε, φαίνονταν διαφορετικό την πρώτη φορά που ψηφίσατε. 07. Υγίτσες και υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 58-83. Υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 58-82. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58-75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58-76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58-88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5877 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 5878 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται άποχες εγκρίνεται Περνάμε τώρα σε 58-58. 58-70, 58-97. Αυτό είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 58-59 και 58-96 ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 89. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται μου φαίνεται, αλλά ας το ελέγξουμε παρακαλώ, την 5889 ηλεκτρονικά. Έναρξη. Πέρασε. 18 υπέρ, 23 κατά, απορρίπτεται. 5891 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται, αλλά δεν είμαι βέβαιος. Έλαχος. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. 24-17. Εγκρίνεται. 68. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 90. Α, όχι. Συγγνώμη, έχει διακρεωθεί. Η 5869 υπέρ. Έναρξη. Πέρας. 20 υπέρ, 21 κατά. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται παρόλα αυτά, ναι. 58-60 και 58-95 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 58-61 71-94-17 όλες μαζί υπέρ κατά άποχες εγκρίνονται 58-62-72-93 ταυτόσιμες υπέρ κατά Άποχες εγκρίνονται. 59-18 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 52-65-87 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 58-66 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59-20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59-23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58-99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος Έναρξη. Πέρας. 17 υπέρ, 25 κατά, μία αποχή. Απορρίπτεται. 59-0-0. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 59-01. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 59-02. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59.03. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59.08. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Πέρας. Ήταν σαφές το αποτέλεσμα, αλλά πραγματικά τον σηκώνει τα χέρια δεν φαίνεται. Αλλά απορρίπτεται, εν πάση περιπτώσει. Ξεκάθαρα. 25, 59, 25, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το ελέγξουμε και αυτό. Την 25 παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. 17 υπέρ, 25 κατά. Απορρίπτεται. 58-79 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59-10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα να περάσουμε στις τροφολογίες στο σχέδιο γνωμοδότηση. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Ας το ελέγξουμε παρακαλώ. Έναρξε. Α, όχι, η τροπολογία 3. Η τροπολογία 3 παρακαλώ ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρασε. 18 υπέρ, 25 κατά απορρίπτεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Ας το ελέγξουμε παρακαλώ. Την 11. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρασε. 20 υπέρ, 24 κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το ελέγξουμε παρακαλώ. Ελέγχουμε τη 14. Πέρας.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 κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για την 28. Πέρας. 22 υπέρ, 21 κατά. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται γιατί είναι 22 υπέρ, 22 κατά μια και ο συνάδελφο δεν έχει την κάρτα του μαζί. Άρα έχουμε ισοψηφία και απορρίπτεται. Αλλά η αποχή ήταν αυτή που καθόρισε το αποτέλεσμα, ξέρετε. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42. Α, καταπίπτει 42. Η 39 εγκρίθηκε. Η 39 την διεκπαιρέωσαμε. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται, μου φαίνεται, ας το ελέγξουμε για να είμαστε βέβαιοι, γιατί 40 παρακαλώ, έναρξη. Πέρας. 25 υπέρ, 18 κατά, έγκρινεται. Και τώρα έχουμε ψηφορές σε τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι να ψηφιστεί το 45 χωρίς ε, την πρόταση αυτή. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται μου φαίνεται. Ας το ελέγξουμε. Έναρξη. Πρώτο τμήμα. Πέρας. 23 υπέρ, 20 κατά. Μία αποχή έγκρινεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 54. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 56. Έλεγχο ζητείται. Μα ήταν σαφές, λέει ο πρόεδρο Το αποτέλεσμα, εν πάση 55 παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Να ελέγξουμε. 20 υπέρ 21 κατά 3 αποχές ήταν οριακό το αποτέλεσμα. Απορρίπτεται ωστόσο. Παρ' όλα αυτά. 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 58. Υπέρ. Κατά αποχές έγκρινεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές έγκρινεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές έγκρινεται. 61 υπέρ, κατά, αποχές έγκρινεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές έγκρινεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές Εγκρίνεται μου φαίνεται. Ας το ελέγξουμε. Έναρξη. Πέρας. 19 υπέρ 25 κατά. Απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Άποχες. Ας την ελέγξουμε παρακαλώ και την 76. Έναρξη ψηφορίας. Πέρας. 21 ψήφι υπέρ, 23 κατά, απορρίπτεται έως εκ τούτου. Και τώρα να περάσουμε στην τελική ψηφοφορία. Έναρξη παρακαλώ. Ο Μάρκος Πίπερ πρέπει να ψηφίσει. Πέρας ψηφορίας. 41 ψήφοι υπέρ, 2 κατά και 1 αποχή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την εισηγήτρια όλος ιδιαίτερος. Έχουμε και άλλες ψηφοφορίες, αλλά δεν είναι τόσο εκτενείς. Σε ό,τι αφορά το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την αποθήκευση φυσικού αερίου, ε, την έκθεση έχει αναλάβει η Κλάουδια Μοντέρο Αγκουάρ Και περνάμε τώρα στη συμβαστική υπερθμόν 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η ένα α συμβαστική υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε παρακαλώ την τροπολογία 11, παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Πέρας. 25 υπέρ, 16 κατά, 2 αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Ας την ελέγξουμε κι αυτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 12. Πέρας. 22 υπέρ, 19 κατά, 2 αποχές. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Προφορική τροπολογία υπαριθμών 1. Είναι κανείς ε, κατά της προφορικής τροπολογία, Όχι. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε παρακαλώ. Για την προφορική τροπολογία ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 20 υπέρ, 23 κατά. Απορρίπτεται. και 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. Τροπολογία 32. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφοφορία σε τμήματα για την 33. Πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε παρακαλώ. Το πρώτο τμήμα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρασε. 19-24 ψήφι, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 34 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε παρακάτω το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 35. Πέρασε. 22 υπέρ, 20 κατά. Εγκρίνεται. Η 36 Υπέρ. Κατά. Αποχέ, συγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. Η 50 παρακαλώ υπέρ. Κατά. απόχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 68 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 79 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 80 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 81 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 82. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 83 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Έλεγχος. Για την 83 παρακαλώ στο τέλεχος. Έναρξη. Πέρας. 23 ψήφοι υπέρ 19 κατά. Σας ευχαριστούμε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται και 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 90 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Αν και μου φαίνεται ότι απορρίπτεται. Την 90 ψηφίζουμε. Έναρξε Πέρας. 27 υπέρ 15 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 91. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 92. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία τώρα. Έναρξη. Πέρας. 37 υπέρ, 38, 5 κατά, καμία αποχή. Εγκρίνεται. Ευχαριστούμε και την εισηγητρία. Και τώρα έχουμε και μία ψηφοφορία ακόμα για τη δεύτερη ανάγνωση, για την ε, θέση του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τα, τις τεχνικές προδιαγραφές για τα πλοία ιστορικής ναυσιπλοείας, κατάργηση της οδηγίας του καθεξής και έχουμε μόνο μία ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Έναρξη παρακαλώ της ψηφοφορίας. Και πέρασε. 40 υπέρ, μία ψήφος κατά, μία αποχή και να συγχαρούμε τον εισηγητή κύριο Μπελέτ και έτσι ολοκληρώθηκαν λοιπόν οι σημερινές ψηφοφορίες. <laughs> well done. Good aber manchmal sieht man wirklich. So, da ein bisschen in Zeitverzug sind, machen wir Και επειδή έχουμε καθυστερήσει λίγο, ας ε, συνεχίσουμε πάρα αυτά. Όσοι δεν έχουν δουλειά, παρακαλώ, εδώ στην αίθουσα, να βγουν γρήγορα από την αίθουσα και να κάνουν ησυχία. Γιατί τώρα θα κοιτάξουμε την έκθεση εφαρμογή σχετικά με την οδηγία του Συμβουλίου για την εφαρμογή τη αρχή τη μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίε και την παροχή αυτών. Ο Γιάννη Νίλσον είναι ο εισηγητή μα και του δίνω παρά αυτό το λόγο. Tack så mycket, herr ordförande. Det här är viktigare för oss än eh, Ευχαριστώ. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, πολύ πιο σημαντικό από ό,τι πολλοί ε, μπορεί να πιστεύουν, γιατί έχει επιπτώσει στις μεταφορές και στον τουρισμό. Και από την εμπειρία μας διαπιστώνουμε και από τη δική μου εμπειρία την ε, τοπική, θα πρέπει να σας πω ότι έχουμε εξετάσει στις περιφέρειές μας ε, τι ευχαριστεί τους, ε, τους τουρίστες και τι ε, όχι. Εδώ και δεκαετίες το, το θέμα της ισότητα είναι, είναι πολύ σημαντικό για τους τουρίστες και γι' αυτό θα πρέπει και να το ε, λάβουμε υπόψη. Υπάρχουν βέβαια κάποια θέματα κλειδιά που πρέπει να εξασφαλίσουμε δηλαδή την ισότιμη μεταχείριση ανδρών και γυναικών ας πούμε όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες αν δούμε για παραδείγματα του ε, sharing economy εκεί βλέπουμε τέτοιες περιπτώσεις αλλά βλέπουμε να υπάρχει και σεξουαλική παρενόχληση στα, μέσα δημόσια, στα δημόσια μέσα μεταφοράς. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ε, Ποιο είναι αρμόδιο όταν τέτοια πράγματα συμβαίνουν, καθώ και να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τις, ε, τα περιστατικά ε, σεξουαλικής παρενόχληση. Οι εθνικές και οι τοπικές αρχές έχουν να παίξουν ρόλο κλειδί στην εφαρμογή αυτής της σημαντικής οδηγία, να κατανοήσουν τα κατημέλη τις υποχρεώσεις τους <coughs> και επίσης πώς θα δοθούν επαρκή σπόροι στις εθνικές αρχές. Τώρα, όσον αφορά την, τον θυλασμό σε δημόσιους χώρους και εδώ ελπίζω ότι οι εθνικές κυβερνήσεις θα καλύψουν ε, αυτήν ε, την ε, πρακτική που είναι πιο σημαντική από ό,τι νομίζουμε. Αυτή είναι η γνωμοδότησή μου και προσβλέπω στις δικές σας παρατηρήσεις για να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο αυτήν την έκθεση. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Σπαχμάν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον συνάδελφο για τη δουλειά που έχει κάνει και όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι το θέμα της ισότητας So, Τώρα λειτουργεί και πάλι το μικρόφωνο μου, λέει ο Ότι το θέμα λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και απασχολεί πολύ κόσμο. Και σε ό,τι αφορά ε, τα θέματα μεταφορών και τουρισμού καλούμαστε να εξετάσουμε αυτά τα θέματα, αλλά υπάρχουν και στην αγορά εργασίας πολλά προβλήματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να πραγματευτούμε εδώ πέρα στην έκταση αυτή. Ο συναδελφός Νίλς ε, σωστά μίλησε για τα προβλήματα στις δημόσιες συγκοινωνίες. Αυτό εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλο πρόβλημα. Και εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε το θέμα της ευθύνη τρίτων. Αυτό το ζητούμε. Ε, και στην ίδια την έκθεση ε, επισημάνθηκε αυτή η ανισορροπία, η ανισότητα που υπάρχει μεταξύ κρατών μέλων, το οποίο και καθιστά την όλη μας εργασία αρκετά δυσχερή. Όλα αυτά λοιπόν εφαρμόζονται με διαφορετικό τρόπο στα διάφορα κρατημέλη και επιπροσθέτως ε, έχουμε και, και διαφορετικά δεδομένα και διαφορετική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε και σωστή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Αυτά λοιπόν ήταν τα σημεία τα οποία θα θέλαμε να αναφέρουμε προσθέτως και να πω τέλος ότι πιστεύω ότι αυτά είναι πολύ σημαντικά και για τον τουρισμό και εδώ ελπίζω να μπορέσουμε να βάλουμε και στο σημείο 6 ε, μία αναφορά στον τουρισμό και κάτι άλλο που λείπει θεωρώ. Αυξάνεται ο αριθμό των γυναικών που οδηγούν λεωφορεία ή φορτηγά και νομίζω ότι έχουμε πολλά προβλήματα σε ό,τι αφορά και τις ε, τοποθεσίες ε, ξεκούρασης και έχουμε προβλήματα συνθήκων υγιεινής και αυτό ασφαλώς και θα απασχολήσει και τις γυναίκες, απασχολείται και τους άντρες να επισημαθεί ίσως και αυτό και κατά τα άλλα πιστεύω ότι η έκθεση είναι πάρα πολύ πλήρης και ισορροπημένη. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Bilbao. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Παίρνω το λόγο για να αντικαταστήσω την κυρία Μέισνερ. Μου έστειλε κάποια λόγια, τα οποία θα ήθελα να σας διαβάσω, γιατί δεν μπορεί να είναι μαζί μας σήμερα στην Επιτροπή μας. Η αντίστοιχη οδηγία υιοθετήθηκε το 2004 Η Επιτροπή υιοθέτησε μία έκθεση χωρίς να αναφέρει τα σχετικά με τις μεταφορές. Είναι διαφορετικές οι τιμές που προσφέρονται σε άνδρες και γυναίκες στην ασφάλιση. Μεταξύ άλλων. Η διάκριση του φίλου λαμβάνει χώρα στην, στις δημόσιες μεταφορές. Στο σημείο 8. Βοήθεια στις εγγύους στα αεροπλάνα. Ή 9. Σεξουαλική παρενόχληση στις δημόσιες συγκοινωνίες. Μπορούν να είναι υπεύθυνοι οι πάροχοι της ε, υπηρεσίας. Θα πρέπει να γίνει συζήτηση. θα πρέπει οι πάροχοι τη υπηρεσία να προλαμβάνουν τέτοιου τους φαινόμενα, να έχουν ειδικού χώρους ε, για τις ε, γυναίκε. Όλα αυτά δεν έχουν επιληθεί. Δεν υπάρχουν ασανσέρ ή άλλα, άλλοι εξοπλισμοί σε όλες τις τάσεις του μετρό ή του τραμ για ε, τους ενδιαφερόμενους, γυναίκες με καροτσάκια, με μικρά παιδιά, άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Θα πρέπει όλα αυτά να ληφθούν υπόψη. Αυτά θα ήθελε η κυρία Μέσνερ να διαβιβάσει και από τη στιγμή που έχω το λόγο κύριε Πρόεδρε να τονίσω δύο θέματα. Καταρχάς, το θέμα των ασφαλιστικών εταιριών. Πράγματι ως γυναίκες υφιστάμενθα διακριτική μεταχείριση διότι έχουμε πιο υψηλά ασφάλιστρα ενώ από την άλλη οι γυναίκες ε, κάνουν λιγότερα ατυχήματα και όταν το κάνουν το ατύχημα είναι λιγότερο σοβαρό. Καλό θα είναι να ρωτωθούμε όλοι γι' αυτά. Έχουν υπάρξει εμπειρίες σε διάφορα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να επιμείνουμε στην κανονικότητα. Μία ευρωπαϊκή χώρα που ξεκινά να καθορίζει το σύστημα δημοσίων μεταφορών προβλέποντας ειδικά βαγόνια για γυναίκες ε, δεν έχει λύσει τα θέματα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης. Υπάρχει ανισότητα και δεν έχει εξαλειφθεί. Θα πρέπει λοιπόν να, η έκθεση να τονίζει όλα αυτά τα ζητήματα και την ανάγκη απαραίτητων έξτρατιών επικοινωνίας και ενημέρωσης για θέματα ισότητας, έτσι ώστε οι γυναίκες που έχουν ευθύνε στις ε, δημόσιες μεταφορές να ε, δουν ότι δεν θα ε, γίνονται θύμα διακρίσεων. Για παράδειγμα, θα έπρεπε ως απαραίτητο η υποδομή να μην έχουμε αλλαξιέρες για τα μωρά μόνο στις τουαλέτες των γυναικών. Σήμερα δεν είναι θέμα μόνο των γυναικών και δεν είναι καν θέμα μόνο των ανδρών γιατί έχουμε και ζευγάρια ιδίου φίλου σήμερα και θα πρέπει όλα αυτά να, να προσαρμόσουμε τις δημόσιες υποδομές στη νέα πραγματικότητα. αλλά και ως προς την ε, άδεια ανατροφής και αυτό δεν θα πρέπει να αφορά μόνο τις, γυναίκας, τις γυναίκες. Σε κάθε περίπτωση, σε κάθε χώρα, μέλη, μέλος πρέπει να γίνει η εκστρατεία ευαισθητοποίησης για να προστατευτούν όχι τόσο οι μητέρες αλλά κυρίως τα παιδιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζιλ έδωσε το λόγο σε δύο άνδρες και γι' αυτό προτίμησα μετά την κυρία Μπιλμπάου. Ο κύριος Ζιλ λέει προτιμώ να μην πω τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα, αυτήν την εβδομάδα έμαθα μια καινούργια λέξη. Γιατί μου πήρε τόσο πολύ, ε, τόσο πολύ καιρό να τη μάθω. Τέλος πάντων, καλό αργά παρά ποτέ. Ανδροκεντρισμός είναι η τακτική, συνειδητή ή μη, του να τοποθετούνται άρενα ανθρώπινα όντα ή μία διάσταση αρσενική ε, οπτικής γωνίας στο επίκεντρο ε, των πεπιθήσεων ε, του ατόμου. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ειδικέ ανάγκες των γυναικών σε θέματα κινητικότητας. Αυτή η τάση προς τον ανδροκεντρισμό είναι κάτι που θα πρέπει να μας ε, βάλει σε επιφυλακή. Φυσικά και το να αλλάζεις ένα μωρό, να θυλάζεις, να σου επιτρέπεται να παίρνεις το αεροπλάνο. Όλα αυτά είναι σημαντικά πράγματα και είναι ε, δράσεις που θα πρέπει να συμπεριλάβουμε, αλλά να μην περιοριστούμε σε αυτές. Οφείλουμε όλοι να αντλήσουμε τα διδάγματα και δεν θα πρέπει να ενδιαφερθούμε μόνο για τον τουρισμό, αλλά για την καλύτερη διαβίωση όλων μας. Όταν έφτασε ένα από τα αυτοκίνητα του Κοινοβουλίου για να με πάει σε μία από τις συσκέψεις του Στρασβουργού, με έκπληξη είδα γυναίκα οδηγό και τη είπα ότι δεν νομίζω ότι με έχει πάρει ποτέ γυναίκα ως οδηγός από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μου εξήγησε ότι από τις 90 οδηγούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μόνο δύο είναι γυναίκες. Επομένως πρέπει πρώτα να ρυθμίσουμε τα του οίκου μας πιστεύω και να αυξήσουμε αυτό τον αριθμό. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει ισότητα των φύλων και στους επιβάτες και στους χρήστες αλλά και στους χειριστές των μέσων μεταφοράς. Είναι ανθρώπινα όντα και αξίζουν το σεβασμό όλων ε, και οι θυλάζουσες γυναίκες φυσικά. Όχι επειδή θυλάζουν, αλλά για όλους ε, τους δυνατούς λόγους. Με αυτό το πνεύμα θα ήθελα να κινηθούμε και να προχωρήσουμε και γι' αυτό θα ήθελα να υποβάλω κάποιες προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιάλα Σέντερ, ευχαριστώ. Χαίρομαι, παρόλο που είναι αργά, ότι, για το γεγονός ότι έχετε ακούσει τη λέξη ανδροκεντρισμός. Ένα φαινόμενο από το οποίο πάσχουμε εδώ και αιώνες. Καλωσορίσατε λοιπόν στο κλαμπ μας των παθόντων από ανδροκεντρισμό. Η χώρα σας είναι μία από τις χώρες που έχει προχωρήσει περισσότερο κύριε Σιγητά ως προς τους κανόνες, ως προς τα μέτρα, ως προς τις εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για ισότιμη πρόσβαση ανδρών και γυναικών στις υπηρεσίες ε, του δημοσίου. Σίγουρα δεν έχετε φτάσει στο 100% αλλά η πρόοδος είναι σημαντική. Η οδηγία μιλά για την πρόσβαση στις υπηρεσίες. Αυτό είναι αληθές. Καταλαβαίνω όμως και θεωρώ ότι οι υπηρεσίες δεν είναι ουδέτερες το πώς παρέχεται η υπηρεσία είναι κάτι που καθορίζεται από τον φορέα αυτό αυτό. Θα ήθελα λοιπόν τρόπον την να είμαστε σε θέση να ενσωματώσουμε συστάσεις ή εντολές για τη ε, δέσμοι της υπηρεσίας, δηλαδή ξενοδοχειακές υπηρεσίες, τουριστικές υπηρεσίες, όλες αυτές αποτελούν ένα πακέτο και ο χρήστης δεν ξέρει ποιος ακριβώς την καθορίζει και πώς την παρέχει αυτή την υπηρεσία, ούτε σε ποια κατάσταση και σε ποιες συνθήκες ζουν και δουλεύουν οι καμαριέρες που καθαρίζουν τα δωμάτια των ξενοδοχείων ή οι μετανάστες που κάνουν τη λάντζα πίσω, ε, στην πίσω αίθουσα του εστιατορίου. Θα πρέπει λοιπόν ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να γνωρίζουν ότι οι υπηρεσίες δεν είναι μόνο ουδέτερες και η ίση μεταχείριση δεν θα πρέπει να είναι μόνο μπροστά στη βιτρίνα αλλά και πίσω, ε, στις πίσω αίθουσες. Ο κύριος Κράμερ έχει πολύ μεγάλη ευαισθησία για τα θέματα αυτά η αρμόδια επίτροπος πριν από κάποιε εβδομάδες, πριν από τις ε, διακοπές του Αυγούστου, οργάνωσε ένα πολύ εντατικό σεμινάριο για τις γυναίκες, για την κινητικότητα και τις μεταφορές. Και ήδη έχουν βγει κάποια συμπεράσματα. Γιατί θεωρώ ότι τα έχει παρουσιάσει ήδη στην ομάδα των φιλελεύθερων. Θα ήταν ενδιαφέρον να έχουμε μια κοινή επιτροπή ή να καλέσουμε την Επίτροπο να μας παρουσιάσει τα συμπεράσματα αυτά. Κάποια από αυτά τα γνωρίζω και άλλοι συνάδελφοι ήταν παρόντες στο σεμινάριο αυτό, όπως και εγώ. Ε, τα πράγματα που λέχθηκαν ήταν πολύ ενδιαφέροντα και νομίζω ότι μπορούμε να μάθουμε πολλά ε, και μας αφορούν όλα αυτά, ειδικά στον τομέα των μεταφορών, στον τομέα της προσφοράς της υπηρεσίας, της παροχής αυτής. Στην Γενική Διεύθυνση για την Έρευνα, όταν καταρτίστηκε ο ορίζοντας για το 2020, καθορίστηκε μια ισχυρή στρατηγική έτσι ώστε όλες οι δράσεις να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη ισότιμης πρόσβασης στην υπηρεσία, στη διαχείριση, στο σχεδιασμό της υπηρεσίας. Ενδιαφέρον θα ήταν να μπορέσουμε να έχουμε συστάσεις προς την Επιτροπή και προς την Επίτροπο και για τα θέματα των μεταφορών. ως προς την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση. Δεν υπάρχει άνεση μεταχείριση μόνο έναντι των γυναικών, αλλά και έναντι των γυναικών με αναπηρία. η διάσταση του φίλου είναι πολύ σημαντική. Έχουμε μητέρες με αναπηρία. Τώρα οι δημόσιες μεταφορές θέλουν να διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση όλων και για λόγους τουρισμού. Αλλά θα πρέπει να μεριμνήσουμε περισσότερο ε, για τις γυναίκες και τα άτομα με αναπηρίες. Ευχαριστώ. Εγώ θέλω να υποστηρίξω αυτή την έκθεση του Γιάνν Νίλσεν. Είναι εξαιρετική και συμφωνώ και με τα σχόλια που έγιναν εξ ονόματο του Άλντε ότι είναι σημαντικό αυτό να διευρυνθεί, να εξετάσουμε δηλαδή ευρύτερα τα θέματα τη φροντίδα. Δεν είναι πάντοτε οι γυναίκε που φροντίζουν, αλλά συχνά οι γυναίκε, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι που βρίσκονται στα μέσα μαζικών μεταφορών είναι, πλήττονται λόγω τη έλλειψη. Ε, ε, προσβασιμότητας πολλές φορές ή λόγω διακρίσεων. Στην Ευρώπη υπάρχουν ε, πολλά προβλήματα. Κάποιες πόλεις θα πάνε πολύ καλύτερα και καλύτερα είναι να προσαρμοστούμε προς το πάνω, προς το καλύτερο. Ε, πιστεύω ότι η Υπηρεσία για την Ισότητα των Φύλων και η Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων του Ευρωκοινοβουλίου ανέδειξαν το ζήτημα. Πρέπει λοιπόν να γίνουν προσπάθειες, γιατί αν οι γυναίκες ιδιαίτερα γνωρίζουν ότι ταξιδεύουν κάπου όπου θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για εκείνες και τις οικογένειές τους να γυρίσουν, ε, μπορεί να είναι φιλικό προς τους τουρίστες, αλλά όχι προς τους ανθρώπους που έχουν δυσκολίε στις τις δημόσιες μεταφορές ή που ταξιδεύουν με μικρά παιδιά ή πιο ηλικιωμένους συγγενείς, τότε σίγουρα είναι δύσκολο να πάνε σε αυτά τα μέρη και αυτό πρέπει να το δούμε συνολικά. Και κάποιες φορές και οι άντρες που ταξιδεύουν με μικρά παιδιά έχουν τα ίδια προβλήματα. Είναι γενικά προς το συμφέρον του κοινού να βελτιώσουμε την κατάσταση για όλους. Αυτό θα τους ωφελήσει όλους, η Κομισιόν. Οικονομική Υπηρεσία τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τους κύριους βουλευτές για τις ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις τους ε, όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας περισσότητας των φύλων στην πρόσβαση αγαθών και υπηρεσιών. Η Κομισιόν θα ήθελε να τονίσει πως όλα τα κράτη-μέλη έχουν λάβει ε, μέτρα για να μεταγράψουν ε, την οδηγία στην ε, εθνική τους νομοθεσία. Ε, η Κομισιόν θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις δραστηριότητες και να στηρίζει τα κρατημέλη ώστε να ε, υλοποιηθεί το πλήρες δυναμικό της οδηγίας και άρα να βελτιωθεί η ισότητα. Δεν θεωρούμε απαραίτητο να προταθούν οδηγίες στην, ε, τροπολογίες στην οδηγία σε αυτή τη φάση, αλλά μπορούμε να συζητήσουμε τα θέματα προσαρμογής, ιδιαίτερα όσον αφορά το πεδίο ε, των εξαιρέσεων που μπορεί να δοθούν. Έχουμε ξεκινήσει δε, δύο διαδικασίες κατά παράβαση και συνεχίζουμε εντατικό διάλογο με άλλα κράτη-μέλη ώστε να εξασφαλίσουμε πλήρη συμμόρφωση προς την οδηγία. Είμαστε απόλυτα δεσμευμένοι να εξασφαλίσουμε την ισότητα σε ολόκληρη την Ένωση και τη σωστή εφαρμογή της οδηγίας αυτής σε όλα τα κράτη-μέλη. Θα λάβουμε βεβαίως υπόψη τις ανησυχίες που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση της ισότητας των φύλων εντός Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα πάλι το λόγο έχει ο συγητής, ο κ. Νίλσεν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Ε, φυσικά και προσβλέπω να, στις ε, ε, οδηγίες, στις τροπολογίες μάλλον που θα υποβάλλετε. Ε, θέλουμε να είναι σύντομη και περιεκτική η δική μας γνωμοδότηση και να περιορίζεται στους δικούς μας τομείς αρμοδιότητας, δηλαδή μεταφορές και τουρισμός. Είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να τονίσουμε περισσότερο τα θέματα του τουρισμού και μπορούμε να βελτιώσουμε την ε, γνωμοδότηση αυτή. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Προθεσμία για την κατάσταση τροπολογίων 8 Σεπτεμβρίου στι 12 το μεσημέρι. Και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο στην ρίζα διατάξη ό,τι αφορά την, ε, το τα διευθυντικά ταμεία και τη μεγιστοποίηση τη αποδοσή του, το λόγο έχει ο εισηγητή, ο κ. Λουτόφσκι. Βελτιστοποίηση τη συμβολή των Ευρωπαϊκών Δραστικών και Παιδικών Ταμείων. Ευχαριστώ και θα μιλήσω πολιτικά. Για να παρουσιάσω τα πιο σημαντικά σημεία τη γνωμοδότησή μα προ την Επιτροπή Ρέτζη τα, την οποία είχα την τιμή να καταρτήσω. Όπως είδαμε και στην προηγούμενη συνεδρίαση, το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι απασχολεί πολλούς από εμάς. Τα πιο βασικά λοιπόν σημεία τα οποία έχετε μπροστά σας αυτή τη στιγμή είναι βεβαίως ότι δεν είναι... Δεν εξαντλούν το θέμα, είναι μια αρχή μόνο της εργασίας μας. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι τα ευρωπαϊκά αντιστατικά ταμεία έχουν συμβάλει σημαντικά στην βελτίωση των υποδομών. Έχουμε διάφορα ταμεία και χάρη αυτά οι μεταφορές αποτελούν πραγματικά τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ωστόσο, δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια και σε ό,τι αφορά τα λάθη που έγιναν και έχουν γίνει κάποια λάθη. Έχουμε κάποια σημαντικά έργα τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί, αλλά έχουμε και κάποια κενά στις υποδομές μας, τα οποία είναι πολύ σαφή στις νοριακές περιοχές και η ολοκλήρωση των έργων TNT δεν θα είναι δυνατή χωρίς την συνέχιση και τη βελτιστοποίηση των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. Το κλειδί λοιπόν για τη σωστή και την επιτυχία είναι ο σωστός προγραμματισμός σε εθνικό επίπεδο αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τις ε, ανάγκες των τοπικών και περιφερειακών ε, επίπεδων. Και θα πρέπει να υπάρχει και καλύτερη λήψη αποφάσεων. Να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει η σωστή εμπειρογνωμοσύνη καθώς και μεταφορά γνώσης προς ε, τα κρατημέλη σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές επενδύσεις. Και επίσης να προσέξουμε όχι τόσο το γεγονό ότι θα πρέπει να αξιοποιούνται τα ταμεία, αλλά ότι οι υποδομέ οι οποίε οικοδομούνται βάσει των ταμείων αυτών θα πρέπει να εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ξέρετε, για τι χώρε τη Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Γιατί αυτό ασφαλώς θα καθορίσει και την εξέλιξη της ευρωπαϊκής μας ενσωμάτωσης. Τώρα, με χαρά θα ακούσω τα σχόλιά σας. Ελπίζω να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη γνωμοτοτήση αυτή και να συμπεριλάβουμε και ενδεχόμενα σημαντικά σημεία τα οποία δεν είχα την ευκαιρία να τα συμπεριλάβω. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρος. Ο κύριος Μοντανκάμπ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο Κοσμά Σλοτοφσκι για το σχέδιο γνωμοδότησης. συμφωνώ ως προς το περιεχόμενο και τα σημεία τα οποία αγγίζει. Μία ερώτηση έχω μόνο και στρέφομαι ενδεχομένω και όπλη στη γραμματεία. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακούμε συχνά αυτό το μότο use it or lose it, ή θα χρησιμοποιήσουμε δηλαδή ένα ταμείο ή θα το χάσουμε. Συμφωνώ, είναι εξαιρετική ως αρχή, αλλά από ό,τι ακούω συχνά, συχνά συμβαίνει αυτό και στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, στις χώρες της συνοχής. Μήπως θα πρέπει να δώσουμε πιο πολύ προσοχή σε αυτό το φαινόμενο. Γιατί είναι κρίμα να έχουμε πόρους για τις ε, υποδομές, για τις μεταφορές και να μην τελικά υλοποιούνται τα προγράμματα αυτά γιατί δεν υπάρχουν άδειε εγκρίσεις, δεν ε, τηρούνται οι προθεσμίες. Και θεωρώ ότι γενικότερα ο προγραμματισμό σε περιφερειακό επίπεδο θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Και επίση δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να εφαρμόζονται με αυστηρέ ε, αρχέ αυτή η αρχή. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, λέει ο πρόεδρο, το use it or lose it δεν είναι θέμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμεί ε, ω κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία το περάσαμε βάσει των εμπειριών που είχαμε συλλέξει σε βάθος χρόνου, που διάφοροι πόροι, διάφορα κονδύλια είχαν περιοριστεί για συγκεκριμένα έργα τα οποία ποτέ δεν υλοποιούνταν. Άρα δεν ήταν δικό τη θέμα της Ευρωπαϊκή Επιτροπής αλλά και δικό μα κυρίω. Η επόμενη εμπειρία. Ε, Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτή τη γνωμοδότηση που πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση, να τονίσω τη σημασία των διαρθρωτικών ταμείων για την εφαρμογή του περιεχομένου του κειμένου αυτού. Θα πρέπει να ενισχυθεί η παράγραφος μεταξύ που τονίζει τις συνέργειες μεταξύ των Ευρωπαϊκών Ταμείων για να έχουμε συνδυασμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για καλύτερη χρηματοδότηση των υποδομών μεταφορών. Δεύτερον, η θεματική συγκέντρωση δεν θα πρέπει να περιορίζει τη δυνατότητα των περιφερειών να επενδύουν στις, ε, στα βιώσιμα μέσα μεταφοράς στις περιφέρειες, στις πιο, περιφέρειες τις πιο ανεπτυγμένες που συχνά δεσμεύονται να εφαρμόσουν συγκεκριμένου θεματικούς άξονες που δεν περιλαμβάνουν τις μεταφορές. Η Επιτροπή να είναι πιο ευέλικτη, να δώσει περιθώριο ευελιξίας στις περιφέρειες. Και τα χρηματοδοτικά εργαλεία υποτίθεται ότι λειτουργούν ως μοχλή, όμως αυτή η λειτουργία είναι πολύ αδύναμη στον τομέα των μεταφόρων. Έχουμε τη διασύνδεση στην Ευρώπη, αυτό το μηχανισμό και οι ενισχύσεις, οι επιδοτήσεις υπό αυτή την έννοια είναι ο καλύτερος τρόπος να χρηματοδοτηθούν οι υποδομές. Έχοντας ακούσει την άποψη διαφόρων περιφερειών, είναι καλό τα διαρθρωτικά ταμεία να μην υπολογιστούν ως κρατικές ενισχύσεις. Και έτσι θα μπορέσουν να υπάρξουν πολύ περισσότεροι φάκελοι, οι τοπικοί παραγόντες να υποβάλουν πολύ περισσότερους φακέλους και να είναι λιγότερο επαχθής και περίπλοκη διαδικασία. Ευχαριστώ. Ο κ. Σας ευχαριστώ. Είμαι σκιώτης εισηγητής εξ ονόματος της Άλτα, αλλά ο βασικός μας εισηγητής, ε, μάλλον σκιώτης εισηγητής δεν μπορεί να προβλεφθεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κι εγώ τον εισηγητή και αυτό το θέμα με απασχολεί ιδιαίτερα γιατί είμαι και σκιώδη στην Επιτροπή ε, Ρέτζι για το θέμα αυτό. Καταρχά να επισημάνω ότι πιστεύω ότι είναι ε, χαμένη ευκαιρία για το γεγονός ότι δεν αναφέρεται τόσο πολύ η κινητικότητα και η αστική κινητικότητα. Θα έπρεπε να αναφέρονται ρητά αυτά ως έννοιες, ε, γιατί σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά δραστικά και τα ταμεία, το θέμα δεν είναι μόνο να υπάρχουν και να δημιουργούνται νέες υποδομές ε, μεταφορών, αλλά και η προώθηση των ε, μεταφορών με χαμηλή εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα, και νομίζω ότι αυτό ισχύει όχι μόνο για την Ανατολική και την Δυτική Ευρώπη, αλλά για όλη την Ευρώπη. Για, γι' αυτό λοιπόν ε, θεωρώ ότι δεν είναι αρμόζουσα αυτή η αναφορά ιδιαίτερα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Οι, τα ευρωπαϊκά διευθυντικά και επενδυτικών ταμείων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παράδειγμα για μια ευφυή ε, κινητικότητα, για ευφυή συστήματα λογιστικής ε, και επιμελητίας, για ευφυείς τρόπους μεταφοράς μέσα στις αυτό θα ήθελα τονιστεί και επιπλέον τα ταμεία αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση κάποιων οικονομικών κλάδων οι οποίοι τώρα συνδέονται με τις ε, μεταφορές αλλά και με τον τουρισμό. Για παράδειγμα και μια στην αυτοκινητοβιομηχανία όπου τα οχήματα του αύριο θα μπορούσαν να οικοδομηθούν με την υποστήριξη των ταμείων αυτών και φυσικά αυτό θα μπορούσε να ισχύει και για τον τουρισμό και αυτό θα ήθελα να τονιστεί πιο πολύ στην έκθεση. Άρα, πρόεδρε, με άλλα λόγια θα καταθέσουμε τροπολογίες και θεωρώ ότι θα υποβάλουμε μια ευρύτατη και πλήρη γνωματότηση στην Επιτροπή Ρέτζη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντέλη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ με τον συνάδελφο Ματής ότι δηλαδή θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να ψηφίζουμε κείμενα με κλιματικούς στόχους, διότι κανονικά το Ευρωκοινοβούλιο όπως και η Κομισιόν θα έπρεπε να μας δίνουν projects τα οποία να κατευθύνονται προς τους στόχους που πρέπει εμείς να συγχρηματοδοτήσουμε. Και όταν κοιτώ τις προτεραιότητες, να θυμίσω ότι κάποια στιγμή πρέπει να κατανοήσουμε πως το σύνολο των ε, προγραμμάτων, όταν μιλάμε ας πούμε, για διεύρυνση αυτοκινητοδρόμων, όπου στην ουσία βολεύουμε τους ε, ε, τις οδικές μεταφορές, ενώ θα πρέπει να επενδύουμε, όπως όλοι το ξέρουμε, στους σιδηροδρόμους. Θα πρέπει λοιπόν να ε, κατευθύνουμε τις μελλοντικέ επενδύσεις για να έχουμε πολυτροπικές ε, μεταφορές, διασυνοριακές μεταφορές, βιώσιμη αστική κινητικότητα. Δεν νομίζω πως μπορούμε να βγούμε από αυτή την έκθεση εάν δεν θέσουμε ερωτήματα για τρεις στόχους. Τους στόχους διοξιδίου του άνθρακα, τους στόχους της ασφάλειας και στη συνέχεια όταν μιλάμε για επενδύσεις, αυτές οι επενδύσεις δεν θα πρέπει να γίνονται παρά μόνο εάν συμβάλλουν ε, τουλάχιστον στην κάλυψη του εξωτερικού κόστους. Σε αυτή την έκθεση λοιπόν το μήνυμα που στέλνουμε είναι να Περάσουμε στον 21ο αιώνα. Δεν πρέπει να ξεκινάμε με τους μεγάλα άχρηστα έργα, αλλά και αστική και βιώσιμη κινητικότητα που δημιουργεί και θέσεις απασχόλησης. Πάντως εγώ από αυτό αναμένω από την έκθεση, σαφές μήνυμα προς την Κομισιόν για αυτά τα ζητήματα και θα ήθελα να προσέχουμε πάρα πολύ, γιατί θεωρώ πως έχουμε να παίξουμε σημαντικό ρόλο ως Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιάλα Σέντερ, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ με τις προτάσεις της ε, έκθεσης. Θέλω μόνο να επιμείνω περισσότερο για το ότι έχουμε πρόβλημα ανάμεσα στα εθνικά προγράμματα και το προγραμματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, εμείς μπορεί να... Και, άρα και με τα, τις κυβερνήσεις. Γιατί αυτή η πρόταση στην ουσία αφορά το Συμβούλιο. Πρόκειται για ένα προγραμματισμό καταπληκτικό, υπέροχο κτλ. Ε, όμως, τα εθνικά προγράμματα δεν συμπίπτουν. Ούτε στα χρονοδιαγράμματα, ούτε στη χρηματοδότηση, ούτε τίποτα. Και αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε ότι πρέπει δηλαδή να εισαχθούν τα θέματα του ευρωπαϊκού προγραμματισμού, τουλάχιστον των ευρωπαϊκών δικτύων, ώστε τα εθνικά προγράμματα να τα λαμβάνουν υπόψη αυτά τα έργα. Που όπως είπα και προηγουμένως δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που συζητάμε σήμερα εδώ, παρότι οι κυβερνήσεις ε, ε, μετέχουν στο Συμβούλιο. Η κατάσταση λοιπόν ε, επιδεινώνεται όσον αφορά την απορρόφηση των ε, κονδυλίων στις χώρες ε, του Νότου. Έχουμε τις δυνατότητες, αλλά επειδή είμαστε κάτω από την πότα της λιτότητας και τα, τις αποφάσεις του κυρίου Κατάινεν, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ήδη προσπαθούμε να φτιάξουμε τον προπολογισμό, ήδη δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να τελειώσουμε τη χρονιά. Έχουμε λοιπόν πρόβλημα στην απορρόφηση. Έπειτα. Έχουμε και πρόβλημα χρονοδιαγράμματος, γιατί με το, τα διάφορα νη συν 1, νη συν 2, νη συν 3 υπάρχει σοβαρό πρόβλημα προγραμματισμού κατασκευής των υποδομών. Λείπει χρόνος αλλά και ε, δυνατότητες μα ε, ακούγαμε, ας πούμε, ότι στη Ρουμανία τα, λογικά κονδύλια ε, να... Ούτε και εκεί όμως τα έχουν καταφέρει. Βλέπουμε ακόμα και στην Γερμανία ε, δημιουργούνται υποχρεώσει ε, ε, εθνικέ τι οποίε δεν μπορούν μετά τα κράτη να τηρήσουν λόγω αυτή τη συμφωνία μεταξύ του και του μη συντονισμού ανάμεσα στα προγράμματα. Θα πρέπει λοιπόν ο προγραμματισμό που οι κυβερνήσει εγκρίνουν για τα διευρωπαϊκά δίκτυα τουλάχιστον να γίνονται σεβαστοί στο όσο αυτός ο προγραμματισμό και στα εθνικά προγράμματα. Ξέρετε λοιπόν πώ γίνεται, το ξέρετε πολύ καλά κύριε Κρέμερ, ότι τα εθνικά προγράμματα δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που εμεί προτείνουμε. Αυτή είναι η δική μα εμπειρία όντω. Ε, το είδαμε και στην ψηφοφορία. Υπήρξε μεγάλη πλειοψηφία για διάφορα έργα και τα κράτη-μέλη ήταν αντίθετα. Και έτσι δεν τα καταφέραμε, γιατί ω Κοινοβούλιο έχουμε χρηματοδότηση μόνο. Και χωρί τι επενδύσει ε, των κρατών μελών, αν δεν υπάρχει επιθυμία και προθυμία, δεν έχουμε κάτι να πετύχουμε, το ξέρουμε, αλλά ε, εν πάση περιπτώσει συμβάλλουμε. Γιατί αν ε, είχαμε 100% χρηματοδότηση θα μπορούσαμε να απαιτήσουμε να ολοκληρωθούν κατά 100% τα έργα. Αλλά εφόσον είμαστε στο 60-70-80% συμμετέχουν και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Χρειαζόμαστε όμως μια καλή συνεργασία και να σας πω ότι ήμουν στην Βαλτική και Εκεί τα ευρωπαϊκά project παίζουν σημαντικό ρόλο και παρόλα αυτά, ε, παρά το γεγονός ότι όλοι συμφωνούν, κάθονται και τσακώνονται για κάποιες μικρολεπτομέρειες και το ξέρω και από περιφέρει στη Γερμανία που εντάσσονται σε διάφορα μοσπονδακρατήδια και μέσα σε μια χώρα ε, μια γραμμή λεωφορείου προκαλεί προβλήματα. Εάν δεν μπορούμε να τα ρυθμίσουμε αυτά σε μια χώρα, τι να κάνουμε. Όσο δεν τα έχουμε καταφέρει λοιπόν εμείς οι ίδιοι, Ας προσέξουμε και να μην κατηγορούμε τους άλλους και να αναφέρω και αυτά που είπε και ο πρώην πρόεδρος της ε, Γερμανίας, Γκούσταμ ε, Χάνιμαν, ότι ε, αν κάποιος κατηγορεί κάποιον άλλον, ενδεχομένω να του γυρίσει μπούμεραν αυτό. Μάλιστα, επόμενος ομιλητής. Thank you very much, Good morning to everybody. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ για αυτή την πολύ ζωντανή και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πολύ χαίρομαι που βλέπω πόσες ιδέες προκύπτουν σε αυτή την Επιτροπή και πόσο διευρυμένοι είναι οι ορίζοντες όλων. Η συζήτηση αποκτά μεγάλη σημασία από τη στιγμή που γίνεται στη δική σας Επιτροπή και από τη στιγμή που επεκτείνεται σε πολλά θέματα που δεν περιέχονται καν στο κείμενο και είναι πολύ πιο φιλόδοξα. Θα ήθελα να τονίσω τρία στοιχεία, αν μου επιτρέπετε. Πρώτον, συνολικό σχέδιο μεταφορών, τα γενικά εθνικά σχέδια μεταφορών αποτελούν μέρος της αιρεσιμότητας εξάντε που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην ιστορία της πολιτικής συνοχής. Μιλούμε για υποχρεωτικές, κανονιστικές, υποχρεωτικά κανονιστικά ρυθμιστικά προαπαιτούμενα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό είναι τρομακτικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι ακριβώς το προαπαιτούμενο κεκτημένο που χρειάζεται για να έχουμε streamlining, ευθυγράμμιση των κονδυλίων να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και μεγαλύτερο αντίκτυπο των ε, κονδυλίων που χρησιμοποιούνται. Υπ' αυτή την έννοια είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι Κάτι που γίνεται κατανοητό σε επίπεδο περιφέρειας. Ισχύει και για τις γενικές μεταφορές πράγματι, τις εθνικές. Και θα μπορέσουμε ενδεχομένως να το διατυπώσουμε με πιο έντονη φρασιολογία. Όπως είπε ήδη και ένα από τα μέλη σας, είναι σημαντικό να επιθυμίσουμε ότι το, η διευκόλυνση, το εργαλείο Connecting Europe, συνδέοντας την Ευρώπη, έχει αναλάβει μεγάλο μέρος ε, αυτού του έργου. Τώρα, ως προς το use or lose, χρησιμοποίησε το ή αλλιώς το χάνεις. Να τονίσουμε τις πτυχές της τεχνικής βοήθειας. Η πολιτική συνοχής παρέχει τεχνική βοήθεια στους δικαιούχους, στις κρατικές αρχές. Μιλούμε για μια καμπύλη μάθησης και η τεχνική βοήθεια έχει ήδη χρησιμοποιηθεί ευρέως από το 2007 γιατί με το στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο είχαμε ένα άλλο εργαλείο ε, βοήθειας για την προσαρμογή και συνεχίζει η εφαρμογή του έτσι ώστε να προετοιμάσουμε τα βαρέα έργα υποδομής, τα μεγάλα έργα υποδομής. Ενδεχομένως ορισμένα κρατημέλη δεν έχουν την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη και εξειδίκευση για να ολοκληρώσουν τα σχετικά έργα. Και το δεύτερο που θα ήθελα να πω σχετίζεται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη στήριξη προς αυτές. Η πρόταση στα κονδύλια, στα ταμεία θα πρέπει να είναι ευκολότερη και θα ήθελα να τονίσω το εγχείρημα απλούστευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε την ομάδα υψηλού επίπεδου για την απλοποίηση και την απλούστευση των διαδικασιών. Έχει δημιουργηθεί αυτή η ομάδα για να ενσωματώσει στις πράξεις μας την εμπειρογνωμοσύνη και την εξειδίκευση που έχει αποκτηθεί επιτόπου, από το ε, δουλειά επιτόπου. για να υπάρχει καλύτερη απορρόφηση και αξιοποίηση ε, των δυνατοτήτων χρηματοδότησης. και να έχουν εκπληρωθεί τα προαπαιτούμενα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Και τώρα πάλι λοιπόν ο εισηγητής για να κλείσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις ε, παρατηρήσεις σας, οι οποίες ήταν όλες πάρα πολύ ενδιαφέρουσες σε ό,τι αφορά τις βιώσιμες ε, μεταφορές και θα ήθελα να αναφέρω επίσης ότι μιας και στην έκθεση αναφέρουμε τη σημασία των ταμείων αυτών για την Ανατολική Ευρώπη. Και αυτό το λέω όχι επειδή είμαι από την Κεντρική Ανατολική Ευρώπη, αλλά επειδή το ξέρω από πρώτο χέρι, ε, προσβλέπω στις τροπολογίες σας. Αλλά παρόλα αυτά θα ήθελα να επισημάνω το εξή. Το έγγραφο αυτό είναι για μια άλλη επιτροπή. Άρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι δεν θα είναι πάρα πολύ εκτενέ. Θα πρέπει ό,τι έχουμε να πούμε να το πούμε συνοπτικά. Σα ευχαριστώ πολύ και με χαρά θα λάβω και τι τροπολογίε Σα ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Ε, λέει ο πρόεδρο. ε, ούκαν το πολλό το F. Μάλιστα. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογίων 12 η ώρα στις 8 ε, Σεπτεμβρίου. Και τώρα ουσιαστικά θα πρέπει να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Δεν έχει έρθει όμω ακόμα η συζήτηση. Σα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Er oh, er Α, κατέφτασε. Μόλι. Α συνεχίσουμε λοιπόν. Okay, wir können jetzt weitermachen. Ας συνεχίσουμε λοιπόν, λέει ο Πρόεδρος, ε, κύριος Φαντανικάμπ. Για καθίστε να συνεχίσουμε. Ο ρόλος του αλλιευτικού τουρισμού στη διαφοροποίηση της αλληλείας. Ήρθαν ο εισηγητής. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt bizottság!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 και θα στέλνουμε λοιπόν την γνωματοδότησή μα στην Επιτροπή Αλληλεία. Κοιτάξτε, εμεί Ουγγροί είμαστε. Περίκλειστο κράτο. Άρα χρειάστηκε πολύ μελέτη της κατάσταση ε, της ελευτικής των χωρών που έχουν θάλασσα. Αλλά ανέλαβα τα καθήκοντα αυτά. Ανέλαβα την γνωματοδότηση αυτή γιατί πιστεύω ότι ο τουρισμός ε, όλο και πιο συχνά αφορά και θέματα αλλίας και πιστεύω ότι πραγματικά έχει πράγματα να πει η Επιτροπή μας, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Υπάρχουν λοιπόν σημαντικά στοιχεία τα οποία και συμπεριληφθήκαν στο κείμενο, γιατί πρόκειται για ένα κλάδο που δημιουργεί θέσεις απασχόλησης Και άλλα σχόλια θα θέλαμε να κάνουμε. προφανώ. ο αλευτικός τουρισμό ε, παίρνει διαφορετικέ μορφέ ε, στι διάφορε χώρε και για παράδειγμα στι χώρε του Μεσογείου παίζει σημαντικό ρόλο. Υπάρχουν λοιπόν αλευτικές δραστηριότητε. Ε. Υπάρχει η αλία αναψυχής. Υπάρχουν και φυσικά μορφές αλίας στα ποτάμια που απαντώνται και στις περικλειστές χώρες. Θα ήθελαμε να τονίσουμε ότι ως ε, Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού της, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να έρθουμε σε επικοινωνία με όλα τα επαγγέλματα που άπτονται τη δραστηριότητα της αυτής. Θέλουμε λοιπόν βιώσιμο τουρισμό ποιοτικό τουρισμό. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο για όλε τι χώρε και θα πρέπει επίση να έχουμε υπόψη μα ότι οι τουρίστε σήμερα είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι και ενήμεροι. Έχουν τα κινητά του, έχουν τι εφαρμογέ του. έχουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίε για κάθε τοποθεσία. Άρα οι μικροί προορισμοί θα πρέπει να προβάλλουν λίγο καλύτερα τον εαυτό του. αν θέλουν να δημιουργήσουν θέσει απασχόληση, αν θέλουν να προσελκύσουν τουρίστε, θα πρέπει να επενδύσουν στην ενημέρωση, στην πληροφόρηση, στην ποιότητα, στον αυθεντικό χαρακτήρα τον οποίο θα πρέπει να προβάλλουν σε μια καλή ισορροπία τιμής ε, και απόδοσης και ήταν ε, πολύ ενδιαφέρον το ότι συνομιλήσαμε και με άτομα που εκπροσωπούν τέτοιες μικρές κοινότητες... ...στις τελευταίε δεκαετίες, ξέρετε, έχουν γίνει πολλές αλλαγέ. Υπάρχουν πολύ μικρές περιοχές που επικεντρώνονταν σε μόνο κάποιες μορφές αλληλείας. Αλλά πλέον έχουν διαφοροποιήσει την ε, προσφορά τους. Ο μαζικός τουρισμός γενικά χάνει το μερίδιο τους ε, στο σύνολό του τουρισμού. Γιατί οι μικρές αυτές περιοχές που είναι έτσι απείραχτες και αυθεντικές ακόμα συγκεντρώνουν πιο πολύ το ενδιαφέρον του κόσμου και των τουριστών. Κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, το υπογραμμίζουμε άλλωστε και στην νομοδότηση. Οι τοπικέ αλληλευτικέ κοινότητε θα πρέπει να διατηρήσουν την ταυτότητά του. Άρα θέλουμε οικοτουρισμό, τουρισμό που θα προστατεύει τι περιοχέ. Ζητήσαμε επίση ε, να απλοποιηθούν κάποιε κατευθυντήριε γραμμέ. Τι σημαίνει λοιπόν ε, οικοτουρισμός Και υπάρχουν και πολλές ε, ε, οργανώσεις που επικεντρώνονται στον τομέα αυτό. Θα θέλαμε λοιπόν να το ε, ερευνήσουμε αυτό. Θα θέλαμε να ζητήσουμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ερευνήσει ποιες είναι οι επιπτώσεις ε, του κάθε τουρισμού στον χερσαίο τουρισμό, στον εσωτερικό τουρισμό. Θα δούμε και τα διάφορα ταμεία που υπάρχουν και πώς θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Και εδώ λοιπόν μιλάμε για τον αλληλευτικό τουρισμό. Υπάρχουν διάφορες, ε, διάφορες τέτοιοι προορισμοί. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας πανευρωπαϊκός διάλογος ε, όπου και οι εκπρόσωποι των λιμένων και οι εκπρόσωποι των αλλιών και οι εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου φυσικά θα μπορούσαν να καθίσουν μαζί για να τα συζητήσουν όλα αυτά. Θα πρέπει να τα προβάλλουμε όλα αυτά και στο διαδίκτυο και να δώσουμε πολύ πιο πολλές πληροφορίες, εφορίες. Να δούμε λοιπόν ε, τους διάφορους προορισμούς ε, για την ε, αλληλεία αναψυχής. Κάτι τελευταίο. Να συμπεριληφθεί μία μικρή, ένα μικρό τμήμα στο Ευρωπαϊκό Κόμβο για τον τουρισμό για την αλληλεία. Αυτά. Αυτά συνοπτικά είχα να σας πω. Ελπίζω να τα κατανοείτε όλοι σας και φυσικά ό,τι ερωτήσεις και παρατηρήσεις έχετε είναι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, δεν είναι εδώ η σκιώτης. Ο κ. Φοντεκάμπ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου το ψάρεμα, λέει ο κ. Γιατί τα φοβάμαι αυτά. Αλλά βαίνει και στο Σχίφενιγκ, ξέρετε, στη Χάγη, στη θάλασσα. Και εκεί είναι μεγάλες και πολλές οι εταιρείε ε, αλίας, αναψυχής. Όπως το είπε ο συνάδελφος, ακριβώς είναι τα πράγματα. Οι αλίες, κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, θέλουν ε, λοιπόν, να προωθήσουν την ε, τουριστική αλία. Γιατί φυσικά υπάρχουν και οι κανονικοί, οι πραγματικοί αλίες, οι οποίοι ασχολούνται μόνο με το ψάρεμα και υπάρχουν και οι άλλοι που θέλουν μια άλλη των δραστηριοτήτων τους και πιστεύω ότι είναι πραγματικά πολύ καλή η γνωμοδότηση που κατήρτισε ο συνάδελφος. Το μόνο που με απασχολεί είναι στο σημείο... Μισό λεπτό να το βρω. Στο σημείο 9 κατά πόσο το Ευρωπαϊκό Ταμείο αλληλευτικών ζητημάτων και Αλίες και ναυτιλιακών ζητημάτων και αλλίες, κατά πόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτές τις τουριστικές δραστηριότητες. Εμείς φυσικά μπορούμε να πούμε ότι θα το θέλαμε αυτό, αλλά να προσέξουμε γιατί σε κάποιες χώρες ε, δυσκολεύεται ιδιαιτέρως ο αλληλευτικός κλάδος και να μην επιβαρυνθεί διπλά από την εξέλιξη αυτή. Και αυτό που ερωτώ είναι κατά πόσον είναι δυνατόν, κατά πόσον περιλαμβάνεται αυτό στην στόχοθεσία και στους στόχους του Ταμείου αυτό. Αυτά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Ζήλια, θα ήθελα να καλωσορίσω και εγώ ξενόματος του εισηγητή μας στην ε, έκθεση αυτή που θα βοηθήσουν όλα αυτά για τη διαφοροποίηση της οικονομίας ε, στις διάφορες περιοχές, θα βοηθήσουν την ανάπτυξη, την καταπολέμηση της ανεργίας κτλ. Ο σκιώδος του ΙΣΙΑΡ τονίζει ότι ένα από τα εμπόδια που αντιμετωπίζει ο αραβικός τουρισμός είναι ότι υπάρχει α, ε, μεγάλη επιβάρυνση με κανονισμούς στην ε, εμπορική ναυσιπλοεία και αυτό οδηγεί σε διάφορα πρότυπα τα οποία δημιουργούν προβλήματα. Επίσης θα πρέπει να προωθήσουμε ένα πανευρωπαϊκό διάλογο μεταξύ των τοπικών ομάδων, των λιμένων, των αλλιέων ε, και των τουριστικών κλάδων. Και θα πρέπει να υπάρξει ε, στενή συνεργασία μεταξύ αλλιέων και τουριστικών κλάδων για να βρεθούν σωστές ε, μορφές επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις και για την διαφοροποίηση της αλίας σε τέτοιες αλλιευτικές περιοχές. Αυτά που αναφέραμε λοιπόν και εμείς. Ότι οι ομάδες δράσης θα πρέπει να συνεργαστούν και θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλίας. Και τέλος, θα ήθελα να πω ότι αυτό που δεν υποστηρίζει ο σκιώδες του ECR είναι ότι θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο EMFF δραστηριότητε ιδιαίτερα για τι γυναίκε. Γι' αυτό λοιπόν εν μέρη δεν ε, το έχουμε θέσει το θέμα αυτό και πιο νωρί. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακόμα μια φορά θα Πάρω το λόγο εξ ονόματος της Μέσνερ που είναι ισκιώδης ε, για αυτή την έκθεση. Για να σας πω λοιπόν ότι η ομάδα ε, Άλντε καλωσορίζει αυτή την πρωτοβουλία για αυτό το θέμα διότι αφορά μια πολύ σημαντική πτυχή που θέλει να ενισχύσει τις τοπικές επιχειρήσεις ε, που χρειάζονται θετική οικονομική όθεση. Ο αλευτικός τουρισμός είναι πολύ σημαντικός για πολλέ πολλές οικογενειακές επιχειρήσεις που εντάσσονται και στο πλαίσιο του περιφερειακού τουρισμού. Πρόκειται για ελκυστικές επιχειρήσεις που μπορούν να συμβάλλουν στην διαχείριση του περιβάλλοντος. Πρόκειται για μια μορφή του τουρισμού δηλαδή που παρουσιάζει νέες δυνατότητες και νέες δυνατότητες για έσοδα. Θα ήθελα να τονίσω δύο σημεία, το σημείο 7 και το σημείο 9 που αναφέρονται στο βασικό στόχο που είναι η πραγματική εφαρμογή. Φαίνεται να υπάρχει μεγάλη ανάγκη και ε, για, ε, μάλλον υπάρχουν πολλές διαφορετικές, ε, διαφορετικοί κανόνες σε εθνικό επίπεδο είναι δηλαδή περίπλοκο και δυσάρεστο για τους αλληλείς να κάνουν πραγματικά το βήμα ε, να μπουν στο τουρισμό. Για παράδειγμα στη Γερμανία υπάρχουν εταιρείε που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον να μετατρέψουν την επιχείρησή τους, αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολο να μετατρέψουν τα σκάφη τους ε, με βάση όλους τους κανονισμούς που ισχύουν. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα του αλληλευτικού ταμείου που πολύ συχνά δεν χρησιμοποιούνται καν για τέτοιου είδους εργασίες ε, μετατροπής των σκαφών για τουριστικούς σκοπούς. Στόχος θα είναι να μπορέσουν οι αλληλείς να ε, μετατρέψουν τις επιχειρήσεις τους. Ε, γι' αυτό και υποστηρίζω τις παραγράφους 21 και 22. Επιπλέον θα πρέπει να δούμε και τον εκπαιδευτικό τομέα στον τουρισμό και αυτά ήθελα να πω για την συνάδελφο Μέσνερ και εγώ ίδια θέλω να ε, κάνω μια παρέμβαση. Συμφωνούμε για την ανάγκη διαφοροποίησης ε, στον τομέα της αλίας, όμως νομίζω πως δεν μπορούμε να να απομακρυνθούμε από τις μεταφορές και τον τουρισμό εδώ. Δεν μπορούμε να χάσουμε το στόχο μας, δηλαδή όσον αφορά το θαλάσσιο ταμείο. Και εγώ είμαι μέρος της, Ευρωπαϊκής, της Επιτροπής Αλληλείας. Όταν μιλάμε λοιπόν εδώ, μιλάμε για ένα τομέα αλληλευτικό τοπικό που έχει μια πολύ ισχυρή ταυτότητα και μάλιστα βρίσκεται σε, σε, συνθήκες να προσφέρει διαφορετικό είδος τουρισμού, περνά από πάρα πολλές σοβαρές δυσκολίες, γιατί, γιατί σε αυτή τη φάση αυτό που λείπει είναι αρκετές ε, ε, ποσοστώσεις για να μπορέσουν να σταθούν ως ε, βιώσιμες και αποδοτικές επιχειρήσεις. Δουλεύουμε πολύ για την βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, για τη διατήρηση των πορών, αλλά έτσι ώστε οι, οι στόλοι που επιθυμούν να εργαστούν στην θάλασσα να έχουν απόδοση εδώ λοιπόν αγγείται το βασικό ερώτημα και οι αντιφάσεις. Όταν ε, μιλάμε για τη χρήση του ταμείου, μιλάμε για τη χρήση του ταμείου από πλευράς εταιριών ή σκαφών που ε, κάνουν αλληλεία. Δεν έχουν αρκετές ποσοστές για να δουλέψουν όλο τον χρόνο και πρέπει να σκεφτούν πώς μπορούν να διαφοροποιηθούν. Κατά τη γνώμη μου, δεν μιλάμε για εταιρείε οι οποίες μπορούν και θέλουν να δημιουργήσουν νέα πράγματα για τομείς για ανθρώπους που δεν ασχολούνται με την αλληλεία παρά μόνο με τον τουρισμό. Ε, γιατί τουλάχιστον αυτοί από την άποψη της αλληλείας θα, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν άλλα κονδύλια να φτιάξουν μια μικρή μεσαία επιχείρηση που θα έχει κεντρική της δραστηριότητα την, ε, τον τουρισμό. Εδώ όμως για αυτό το, τα, κονδύλια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε αυτή την πτυχή ότι είναι αλληλευτικές επιχειρήσεις που κοιτάνε να διαφοροποιηθούν. Πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε στον τομέα τον αλληλευτικό, στα σκάφη και τους αλληλείς που λόγω της περίπλοκης πραγματικότητας, κυρίως λόγω της έλλειψης ποσοστώσεων, περνάνε πάρα πολύ δύσκολες ώρες και αναγκάζονται να στραφούν αλλούν. Χρειάζονται, χρειάζονται ε, κονδύλια γιατί δεν είναι εύκολο ένα αλληλευτικό σκάφος που μπορεί να αλληλεύει τρει μήνες μόνο το χρόνο. Δεν είναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί και για να αλλιεύει άλλου είδους ε, ψάρια και να μεταφέρει και επιβάτες τουρίστες. Πρέπει λοιπόν να δούμε και η ενημέρωση είναι... Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ε, τις δυνατότητες αποδοτικότητας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ένα τομέα που πρέπει να ζήσει από αυτή, από αυτή την ιστορία μέσα στο συμμετοχή των γυναικών, ε, θα, ε, σε όλη αυτή την υπόθεση θα πρέπει να δούμε και τη συμμετοχή των γυναικών, που είναι αυτές που επέτρεψαν τη διατήρηση αυτού του τομέα σε πάρα πολλές ακτές του τομέα. Και θα πρέπει λοιπόν να ε, ασχοληθούμε και με αυτή την υπόθεση. Επίσης να μιλήσουμε και για το τι ακριβώς είναι η, ε, αλληλεία αναψυχής και τα σκάφη αναψυχής ξεπερνούν σε πολλούς δήμους τα αλληλευτικά σκάφη με τη δυνατότητα να αλλιεύουν για αναψυχή και θα πρέπει να αναλύσουμε τον αντίκτυπο που έχει αυτή η αλληλεία η, η, αναψυχής επί της επαγγελματικής αλληλείας. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί, όπως σας είπα, να ξεπεράσουν τις ποσοστώσεις και πώς μπορούμε όλα αυτά να τα συμβιβάσουμε. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση λοιπόν για την ανάπτυξη του, της τουριστικής αλίας και κυρίως ε, όσον αφορά τη βοήθεια και την ανάπτυξη της αλληλείας της ίδιας. Ευχαριστώ. Η κυρία Κάρη Μαντελή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματι ε, της ε, σκιώδους μας της κυρίας Εύανς ε, ε, που δεν μπορούσε να είναι παρούσα σήμερα και η οποία θέλει να σας συγχαρεί για αυτή την πρώτη έκθεση. Ωστόσο έχει να εκφράσει και πολύ... έχει να ε, συνομιλήσει να μιλήσει για το ότι ο αλληλευτικός τουρισμός θα πρέπει ε, βασικά να γίνεται με βάση την προστασία της φύσης, του φυσικού περιβάλλοντος και της φυσικής κληρονομίας. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι μας κατεβαίνει με τη φύση πλέον. Ε, και άρα αυτός είναι ο πόρος για τον τομέα του βιώσιμου τουρισμού, ενός τουρισμού που συνδέεται με την αλληλεία και που θα πρέπει στενά να συνδέεται με τα συμφέροντα των μικρών ε, των μικρών βιοτεχνικών δραστηριοτήτων ε, για να δούμε ακριβώς ποιες είναι οι ανάγκες και ποιες είναι και είναι τα μέτρα που θα πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή για να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας. Δεύτερο σημαντικό σημείο είναι αυτό το θέμα που είναι σημαντικό, όπως σας, ναι, συμφωνούμε, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε όλες τις, ε, ελεκτικούς που είναι στις ακτές και τα νησιά και στις λίμνες και στα ποτάμια. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά για να μπορέσουμε μετά να τα προσαρμόσουμε. Σας ευχαριστώ. Äh, Σας ευχαριστώ. Σουίτσα του Μπραφκα. Äh, želim pozdraviti ovo izvješće i kao izvjestiteljica u Sjeni uglavnom se να καλωσορίσω λοιπόν την έκθεση αυτή ως κοιόντας ε, ε, σύμφωνο με το κείμενο και πιστεύω ότι είναι σημαντική η σχέση μεταξύ της αλληλείας και του τουρισμού. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις μικρές αλλαυτικές κοινότητες. Ε, εγώ είμαι στον Ντουμπροβνίκα, από τον Ντουμπροβνίκα έρχομαι, ε, που είναι στην ακτή. Και πιστεύω λοιπόν ότι πραγματικά είναι πολύ σημαντικό το σκέλος του της Αλίας για την ανάπτυξη του τοπικού και του περιφερειακού τουρισμού. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της Κροατίας για την ε, ένταξη στην Ένωση, αποδεχτήκαμε κάποια πρότυπα τα οποία δεν βοηθούν τόσο τις τοπικές κοινότητες. Ελπίζουμε με την πάρτα του χρόνου και με την έκθεση αυτή εν μέρει να καταφέρουμε να αλλάξουμε κάποιους από τους ε, κανονισμούς που υπονομεύουν την αλληλεία και την ταυτότητα την ίδια των τοπικών κοινοτήτων δεδομένου δε του ότι κάποιες ε, τέτοιες κοινότητες ε, ζουν αποκλειστικά και μόνο από την αλληλεία. Η πολιτισμική λοιπόν κληρονομιά θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα σε ό,τι αφορά τη διατήρηση της ταυτότητας των τοπικών κοινοτήτων. Και ένας τρόπος που καθορίζεται και ο χαρακτήρας των, των κοινοτήτων αυτών είναι και η αλία. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε λοιπόν την ύπαρξη των μικρών αλλιών. Και η προσαρμογή των αλευτικών σκαφών, των μικρών αλευτικών σκαφών δεν θα είναι κάτι το απλό, ξέρετε, γιατί πολλοί τουρίστες θέλουν να να πηγαίνουν σε τέτοιους μικρούς ε, προορισμούς. Αυτό γίνεται όλο και πιο δημοφιλές. Ε. Και ελπίζω λοιπόν ότι η έκθεση αυτή, η γνωμοδότηση αυτή τελικά θα καταστεί αποδεκτή με κάποιες μικρές τροπολογίες που θα προτείνουμε. Σας ευχαριστώ από την ε, Κομισιόν, κυρία Γκένοβα, παρακαλώ. Αξιότιμα μέλη, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Όπως γνωρίζει η Επιτροπή σας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναφέρει ότι ο θαλάσσιος τουρισμός είναι ένας από τους τομείς για ανάπτυξη, ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός. Και γι' αυτό έχουμε καταρτήσει μια στρατηγική που εντοπίζει τους στόχους και παρουσιάζει δράσεις που πρέπει να αναλάβουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Μία από, από αυτές τις δράσεις καλή για τη διαφοροποίηση του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού υπό τον άξονα της βιωσιμότητας και της σωστής διαμόρφωσης του τουριστικού προϊόντος. Έχουμε διάφορα έργα διεθνικά με διάφορους θεματικούς, θεματικούς άξονες για τους δρόμους της Ευρώπης. Θέλουμε να συνδέσουμε την αλία με τον τουρισμό και θέλουμε να έχουμε κοινή, να υπάρχει κοινή διαχείριση, η από κοινού διαχείριση με τα κράτη-μέλη και τους τοπικούς παραγόντες ανάπτυξης. Την προηγούμενη εφαρμοστική περίοδο 2007-2013 έχει γίνει η προπαρασκευαστική δουλειά πάνω από 300 τοπικές ομάδες αλλιευτικής δράσης έχουν ε, δημιουργηθεί το 80% αυτών εντόπισαν δράση σε σχέση με τον τουρισμό και τις θεώρησαν ως βασική προτεραιότητα. Βασικός στόχος είναι να ενθαρρύνει τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων, να αυξηθεί το εισόδημα των αλλιέων και να εμπλακούν σε δράσεις συμπληρωματικότητας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην περιβαλλοντική αηφορία των πόρων. Και γι' αυτό χρηματοδοτούνται ε, προγράμματα και έργα που προσθέτουν στο τοπικό προϊόν που συνδέουν την αλληλεία με τη γεωργία ε, και την ε, ενίσχυση του αλληλευτικού τουρισμού πάντοτε σε συνθήκες αηφορίας και βιωσιμότητες. Το άρθρο 13 δίνει τη δυνατότητα στους αλληλείς να υποβάλουν αίτηση για οικονομική στήριξη για ε, ε, επισκευή του αλευτικού σκάφους και μετατροπή αυτού σε σκάφους που εξυπηρετεί τουριστικούς σκοπούς για λόγους τουρισμού. Το κράτος μέλος μπορεί να επιλέξει να τύχει αυτή τη στήριξη ή όχι. Και υπάρχει άρθρο επίσης που προβλέπει τη δυνατότητα στήριξης για την κατάρτιση και εκπαίδευση των νέων αλλιέων. Τώρα, Για το σημείο 11 και για την ανάγκη ανάλυσης οικονομικού αντικτύπου για την ψυχαγωγική αλληλεία υπάρχουν μέτρα για την προώθηση της διαφοροποίησης. Και έχουμε και υδατοκαλλιέργεια στην Εδοχώρα. Έχουμε συνεχή αξιολόγηση και έτσι θα καταλάβουμε καλύτερα τον αντίκτυπο αυτών των μέτρων. Για το 11 και το 18 λέμε ότι η αποτελεσματικότητα της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντική γιατί το 2014 υπήρξε μια μελέτη που με αξιολόγησε τον αντίκτυπο στην τοπική αλλιευτική κοινότητα. Ανατέθηκε η μελέτη αυτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα πορίσματα είναι ότι 5.500 έργα ε, ε, έγιναν το 2013 στηρίζοντας τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στον τομέα της αλίας και μπορείτε και να τη δείτε και στο διαδίκτυο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αλλιευτικών Περιοχών, το FARNET, αξιοποιεί το, τη σύνδεση μεταξύ βιώσιμου τουρισμού και διαφοροποίησης της αλληλευτικής δράσης. Το δίκτυο αυτό το Farnet, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αλληλευτικών Περιοχών, θα οργανώσει συσκέψεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ ηθινόντων του τουρισμού, εκπροσώπων των αλλιέων και των τοπικών αρχών. Η συνεργασία μας στο σημείο 20 είναι σημαντική. Ε, ίσως ε, οι συνάδελφοι από την άλλη Γενική Διευθύνση θέλουν να πάρουν το λόγο και να προσθέσουν κάτι επ' αυτού. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τον εισηγητή και την Επιτροπή σας. Περιμένουμε τα σχόλιά σας για τη βελτίωση του, του, της τουριστικής δραστηριότητας και του αληφτικού τουρισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ χρήσιμα όλα αυτά τα σχόλια που ακούστηκαν. Κάποια ήδη τα έχουμε βάλει στο κείμενο, κάποια άλλα θα τα βάλουμε αργότερα. Σε κάθε περίπτωση ελπίζω να είμαι, είμαστε σε θέση να ε, ικανοποιήσουμε όλους τους ε, συμμετέχοντες, όλους όσοι έχουν συνεισφέρει με σχόλια. Το έχουμε ήδη πει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμφωνεί. Αν υπάρχει κάποιο σχόλιο καθυστερημένο θα το περιμένουμε και μετά θα υποβάλουμε την έκθεση. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ όλους. Σας ευχαριστώ. 13 Σεπτεμβρίου, 12 η ώρα το μεσημέρι, προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών. Και τώρα να περάσουμε στο επόμενο σημείο στην ημερήξη διάταξη. Είναι η κρίση και η υποπτή τη αγορά των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ορμονικού του και των συστημάτων κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών των μονάδων που προορίζονται τα οχήματα αυτά. Κάριμα Δελή, η εισηγήτρια. Ε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λυπούμε διότι δεν έμειναν οι συνάδελφοι να ακούσουν για αυτό το θέμα το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αγαπητοί συνάδελφοι, η γνωμοδότηση που θα εγκρίνουμε τον επόμενο Νοέμβριο για την υποδοχή και την επιτήρηση των αγορών οχημάτων είναι ουσιοδότηση ουσιώδους σημασίας και επιμένω στο χαρακτηρισμό ουσιώδους γιατί έχουμε ένα κανονισμό που θα έχει ένα τεράστιο αντίκτυπο στην αυτοκίνητο βιομηχανία και ελπίζουμε και το επιθυμώ εγώ σφόδρα να έχει θετικό αντίκτυπο στην υγεία μας, στο κλίμα μας και στην ασφάλειά μας και θα είμαι ξεκάθαρη και σαφέστατε μετά το σκάνδαλο Volkswagen Ζήτησα από την ομάδα μου τη σύσταση ερευνητικής και εξετιστικής επιτροπής. Χαίρομαι που οι άλλες ομάδες οι πολιτικές την στήριξαν και υπάρχει αυτή η διερευνητική επιτροπή και όσοι συμμετέχουν και πολλοί από εμά συμμετέχουν σε αυτή τη διερευνητική επιτροπή γνωρίζουν πόσο επικοδομητικά διδασκόμαστε μαθήματα από την παρουσία μας στη διερευνητική αυτή επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέτρεψε να διωγγωθεί ένα σύστημα όπου η απάτη είναι δυνατή, όπου βελτιστοποιούνται οι δυνατότητες των αυτοκινήτων με νόμιμο τρόπο να υπάρχουν αποκλήσεις μεταξύ εργαστηρίου και πράξης ε, ε, σε ό,τι αφορά τις εκπομπές των διαφόρων αερίων που είναι 10 φορές τελικά ε, υψηλότερες από τον κανόνα και από τα πρότυπα. Τα αποτελέσματα αυτά έχουν επιβεβαιωθεί από εθνικές επιτροπές που έχουν συσταθεί σε διάφορα κρατημέλη και όλοι καταλήγουν καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. Τα πρωτόκολλά μας πιστοποίησης και ελέγχου δεν κάνουν. Δεν είναι καλά. Ε, τίθεται η κυκλοφορία αυτοκίνητα στην Ευρώπη. Υποτίθεται ότι έχουν περάσει τα τεστ για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και άλλων αερίων και πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και λαμβάνουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης και το καθεξής. Όμως δεν τηρούν τελικά τους κανόνες παρά μόνο με, ε, στα πρώτα χιλιόμετρα που διανύουν και όχι στα επόμενα. Και είναι ειδική ευθύνη της Επιτροπής εμείς να τα αναδείξει όλα αυτά. Αφήσαμε να εδρεωθεί ένα σύστημα το οποίο είναι εις βάρος του γενικού ευρωπαϊκού συμφέροντος. Και τι εννοώ με τη λέξη σύστημα. Θα σας δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα για να το περιγράψω. Σήμερα το σκάνδαλο Volkswagen έχει δείξει ότι υπάρχουν μηχανισμοί ακύρωσης παράνομης ή μάλλον παράνομης επικύρωσης, αλλά και νόμιμης. Βάσει του κανονισμού 715 του 2007. Μπορεί δηλαδή κανείς να επενεργοποιήσει αυτό το πράγμα τη στιγμή που το αυτοκίνητο περνάει το τεστ και μετά να το ξαναθέσει σε ισχύ και να το ενεργοποιήσει. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε τέτοιε πρακτικέ. Στι ΗΠΑ, στι ΗΠΑ δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, δεν γίνονται. Εξού και έχουμε τις τεράστιες αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών συνθήκων οδήγησης και των συνθήκων εργαστηρίου. Και χρειάστηκε να περιμένουμε το 2017 να έρθει με τη θέση σε ισχύ των νέων προτύπων έτσι ώστε να καταλάβουμε ότι για τα μέτρα εκπομπών πρέπει να μπει ανιχνευτής στην εξάτμιση. Τόσα χρόνια, τόση αδράνεια, ε, είναι συστημική αδράνεια αυτή, μέρος του συστήματος λοιπόν. Και τελικά οι ψηφοφόροι, οι πολίτες ε, και άρα οι καταναλωτές, ε, τι τους λέμε θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αγοράζει κανείς ένα όχημα το οποίο βάσει των ε, τεστ ε, καταναλώνει π.χ. 6 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα. Από την πρώτη φορά που θα το γεμίσετε συνειδητοποιείτε ότι καταναλώνει 20 ή 40 φορές περισσότερο και από αυτό που είχατε διαβάσει στο φυλάδιο και θεωρείτε ότι είναι φυσιολογικό. Όχι, δεν είναι φυσιολογικό και δεν μπορούμε να το ανεχθούμε. Να υπάρχουν τέτοιου είδους υπερβάσεις. Γιατί οι ρηπογόνες αυτές εκπομπές 20 φορές περισσότερο από τα τεστ οδηγούν σε προώρους θανάτους κατά δεκάδες χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδες Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, 70.000 είναι οι πρόοροι θάνατοι λόγω της ατμοσφαιρικής ρήπασης, που οφείλεται κατά κύριο λόγο σε τέτοιου είδους εκπομπές. Περιμένουν οι πολίτες να τους εγγυηθούμε ότι η ποιότητα του αέρα θα βελτιωθεί. Δεν χρησιμεύει σε τίποτα και δεν έχει κανένα νόημα να θεσπίζουμε κανόνες και να έχουμε ε, τον πύχη ψηλά Euro 5, Euro 6, ε, για τις εκπομπές μονοξυδίου του άνθρακα και ούτω καθεξής, εάν δεν έχουμε παράλληλα ένα συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο που να επιτρέπει στη βιομηχανία να τηρεί αυτά τα πρότυπα και αυτούς τους κανόνες. Οι πολίτες περιμένουν από εμά να είμαστε ανεξάρτητοι και να έχουμε διαφάνεια σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Περιμένουν από εμά να έχουμε ένα νέο σύστημα εποπτείας και επιθεώρησης των αγορών που να λειτουργεί, που να είναι αποδοτικό. Δεν υπάρχει σήμερα και θα το θεσπίσουμε να έχουμε τακτικό έλεγχο καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του οχήματος, όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ για παράδειγμα. Οι πολίτες περιμένουν από εμά να αναλάβουμε δράση για να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη τους στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η έκθεσή μου δεν έχει σκοπό να λειτουργήσει ως αστυνόμευση των κατασκευαστών και των αυτοκινητοβιομηχανιών. Αυτός ο ρόλος είναι για την Επιτροπή ΕΜΙΣ. Οι δήμαρχοι των μεγάλων πόλεων έχουν προσφύγει στο δικαστήριο ε, και έχουν συνέργεια. Εγώ υποβάλλω προτάσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών ελέγχου και τη βελτίωση του καθεστώτος κυρώσεων για να έχουμε αυτοκινητοβιομηχανία αξιόπιστη επιτέλους. Στην έκθεση λοιπόν έχω διάφορες ομάδες τροπολογιών. Πρώτον, τροπολογίες με σκοπό να μειωθεί σημαντικά ο κίνδυνος ενός νέου gate. Δημιουργείται μια Ευρωπαϊκή Αρχή Εποπτείας, Επιθεώρησης, ανεξάρτητη, που μπορεί να κάνει τα δικά της τεστ και τις δικές της ε, ε, δοκιμές, όπως έχουν και οι Αμερικάνοι τη δική τους προστασία, ε, υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος. Προτείνω τη σύσταση, την επιβολή συστημάτων σου κυρώσεων. Ίδιο παντού στην Ευρώπη με αντισταθμίσεις, με αποζημιώσεις, με, με, με, το οποίο να ισχύει και να εφαρμόζεται ε, παντού. Δεύτερη ομάδα τροπολογιών για την ε, επικύρωση των οχημάτων. Πρέπει να ενερμονίσουμε, να ξεκαθαρίσουμε το ρόλο των αυτοκινητοβιομηχανιών, των τεχνικών υπηρεσιών και των εθνικών αρχών. Δεν έχουν διαιρεθεί ξεκάθαρα αυτοί οι ρόλοι σε όλες τις χώρες. Δεν υπάρχει ξεκάθαρος διαχωρισμός και κατανομή των ρόλων του δημοσίου και του ιδιωτικού, το τι κάνει ο καθένας και πρέπει να έχουμε ανεξαρτησία και διαφάνεια μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Τρίτη ομάδα τροπολογιών για την εποπτεία και επιθεώρηση των αγορών. Μια ευρωπαϊκή αρχή με δικό της προϋπολογισμό, με πραγματικές εξουσίες, να μπορούν τουλάχιστον να απαιτούν από τις εθνικές αρχές να ανακαλούν τα οχήματα για τα οποία υπάρχει υποψία ότι ε, είναι ανεπαρκή και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Σας καλώ λοιπόν να υπάρξει ένα δεύτερο κύμα τροπολογιών. Πρόσεξα ιδιαίτερο τα απορίσματα της Διερευνητικής Επιτροπής και των Εξεταστικών Επιτροπών, όλων αυτών των επιτροπών που έχουν ερευνήσει το θέμα στις διάφορες χώρες και κυρίως στη Γαλλία. Και τα απορίσματα, τα συμπεράσματα, οι συστάσεις για ορισμένες που προκύπτουν από ορισμένες εκθέσεις, κυρίως γαλλικές, μας ήρθαν στο κείμενο το καλοκαίρι, μας ήρθαν το καλοκαίρι, δεν μπορέσαμε να τις βάλουμε στο κείμενο, αλλά πραγματικά πρέπει να έχουμε τροπολογίες για να τις περιλάβουμε. Να περιλάβουμε αυτά τα απορίσματα. Υποχρεωτική πρόσβαση στο λογισμικό του οχήματος, στο software, τη στιγμή του ελέγχου για παράδειγμα, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε του κατά πόσο υπάρχει το παράνομο λογιστικό που ε, κρύβει, που λειτουργεί σαν μάσκα τη στιγμή που το όχημα περνάει τον έλεγχο ή όχι. Κύριε Πρόεδρε, ε, μακρηγόρησα λίγο, ξεπέρασα τα πέντε λεπτά. Θεωρώ όμως ότι αυτή η έκθεση λεπτα θεωρω ομω οτι αυτη η εκθεση πρεπει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, στο ύψος των προσδοκιών των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο θα έπρεπε κανονικά να πάρει ο κύριο Κούνα, αλλά μιας και ο κύριος ε, Σίλια να... Μάλλον επειδή έπρεπε να μεταβεί σε άλλη επιτροπή, το λόγο θα πάρει ο κύριος Ζήλια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξ ονόματος του κύριου Βεσενόφσκη, που ήταν ο εισηγητής, ο δικός μας και ο μάλλον για αυτή την έκθεση, θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει ευρύτερο ρόλο ε, στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Δυστυχώς το Dieselgate έβαλε σε, δύσκολες, ε, ε, σε δύσκολη περίοδο όλη την αυτοκινητοβιομηχανία. Εμείς θα πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε έναν ισορροπημένο τρόπο να προσεγγίσουμε την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Η πρόταση της Κομισιόν δημιουργεί ένα νέο επίπεδο ελέγχου που κατά τη γνώμη μας προσθέτει νέα φόρτιο και υποβαθμίζει το ρόλο των κρατικών αρχών όπως η έκθεση, η, μάλλον ο έλεγχος μέσω του type approval, της έγκρισης τύπου από τις αρχές των κρατών. Δεν στηρίζεται ωστόσο, ε, δεν στηρίζουμε την νέα υπηρεσία, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εποπτείας για την αυτοκινητοβιομηχανία όπως προτείνει ο εισηγητής, ωστόσο θα υποβάλουμε τροπολογίες και προσβλέπουμε στις ε, διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους σκιώδεις. Ευχαριστώ. Ο Βέρνερ Κούντ, σας ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό, το οποίο αφορά το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας και ασφαλώς τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και τα θέματα υγείας των πολιτών. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν περιοριζόμαστε μόνο στις εκπομπές όμως αυτές, Και η κυρία Νταλή φέρνει κάποιο τμήμα τη Επιτροπή εμεί στα πλαίσια εδώ πέρα τη δική μα Επιτροπή. Αλλά αυτό είναι ένα τμήμα μόνο. Σε ό,τι αφορά την έγκριση και υποπτία τη αγορά των μηχανοκινητών οχημάτων και των εμπολικουμένων του, αν θα πρέπει όλα αυτά να ληφθούν υπόψη και οι 400 σελίδε όλων των προσαρτημάτων επίση, ε, διαπιστώνουμε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ ε, συγκεκριμένα, γιατί μιλάμε και για τα αρμουλκούμενα, τα δεν επηρεάζονται από τις ε, ε, προδιαγραφές για τι ε, εκπομπές, εκτός πια και αν είναι τόσο κακοφτιαγμένε που χρειάζεται κατάλληλο περισσότερο καύσιμο για να μπορούν να ρημουλκηθούν. Για να απαντήσω σε αυτά που είπε η κυρία Ντελή, είναι απαραίτητα απαραίτητο οι αρχές για την έγκριση των οχημάτων να εφαρμόζουν τα ίδια εργαλεία και μέσα. Τονίζουμε εδώ και υπογραμμίζουμε τη διαφάνεια και εδώ χρειαζόμαστε αφενός ε, έναν ε, ανεξάρτητο ελεγκτή, μια ελεκτική εταιρεία η οποία θα επιβεβαιώσει το τι έχει συμπεριληφθεί στο όχημα, το έχει να κάνει αυτό με την ε, οδήγηση, με το ηλεκτρονικό σύστημα οδήγησης ε, και καταμέτρηση και κατά να υπάρχει υπάρξει κάποια νοθεία εκεί. Όλα αυτά λοιπόν είναι απαραίτητα να υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα του παραγωγού. Το ίδιο πρόβλημα είχαμε και με το PTI τότε. Ποιος αποφασίζει τελικά και ποιος ε, τελικά αποκαλύπτει τι συστήματα χρησιμοποιούνται και ποιος αποφασίζει ποια εγκρίνονται και πια όχι. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να βρούμε μια ρύθμιση η οποία θα διτεθεί μετά στις εθνικές αρχές προκειμένου να μπορέσουν και αυτές να κάνουν τους ελέγχους τους. Και νομίζω ότι μια τέτοια έγκριση τύπου δεν θα πρέπει να είναι και κάτι μόνιμο. Θα πρέπει να επαναλαμβάνετε και τονίζω ότι χρειαζόμαστε διαφάνεια. Real drive emissions, ε, πραγματικές εκπομπές, ε, εδώ φυσικά δεν χωράει αμφιβολία. Χρειαζόμαστε ίδια κριτήρια σε όλη την Ευρώπη. Και συντονισμό και συνεργασία των τεχνικών υπηρεσιών είναι πάρα πολύ ωφέλιμο. Έω τώρα υπεύθυνη για την εποπτεία αυτή ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήθελε σε κάθε περίπτωση να την κρατήσει Νομίζω ότι θα είναι ε, πολύ ε, έντονες συζητήσεις για το κατά πόσο χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή εποπτική αρχή. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, αλλά ο αυστηρό διαχωρισμός των ε, αυτοκινητοβιομηχάνων και της τεχνικής υπηρεσίας και της υπηρεσίας έγκρισης είναι κάτι το εντελώς απαραίτητο για να μην υπάρχουν παρανοήσεις. Είπε η κυρία Τελή ότι θα πρέπει να υπάρχουν ενιαίες δομές εφαρμογής τελών. Αυτό ναι. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορούσε πραγματικά σε όλη την Ευρώπη να οριστεί ένα ενιαίο επίπεδο τελών. Αυτό πιστεύω ότι θα αποτελούσε πρόβλημα. Αυτό που είναι πολύ απλά σημαντικό είναι ότι στο ιστορικό της Ευρώπης θα πρέπει να έχουμε ίσους όρους για την ε, κατασκευή οχημάτων τεχνικής έγκρισης, τεχνικής αδειοδότησης και τέλος να υπάρχει real drive situation, όχι μόνο δηλαδή για τις εκπομπές, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα ανταλλακτικά και τμήματα. Χαίρομαι ιδιαίτερα και προσβλέπω στη συζήτηση με την κυρία Ντελή. Όσοι θα πάει και στον τριμερή διάλογο. Μιλήσαμε και για την διαφάνεια, ελπίζουμε να προσκληθούν και οι σκιώδεις. Λοιπόν, όταν θα συζητήσουμε τα τεχνικά ζητήματα, κάποιοι από τις άλλες, ε, ε, κάποιοι άλλοι συνάδελφοι από άλλες ομάδες είπαν ότι ενδεχομένω να χρειάζεται να περιμένουμε πρώτη την εκθεσία. Εμείς εγώ πιστεύω ότι το χρειάζεται, γιατί δεν έχει να κάνει το ένα με το άλλο. Θα έχουμε κάποια διάμεσα αποτελέσματα τα οποία θα τα δημοσιεύσει η Επιτροπή. εμεί θα τα δημοσιεύσουμε κι εμεί, αλλά πρέπει να δράσουμε άμεσα, γιατί καθημερινά ε, δίδονται εγκρίσει σε εκατοντάδε καινούργια οχήματα στην Ευρώπη. Θα πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση λοιπόν και real drive emissions προκειμένου να μην ξεσπάνε σκάνδαλα όπως το τελευταίο. Ευχαριστώ. Merci. Effectivement... Ευχαριστώ. Πράγματι, είναι πολύ επίκαιρο θέμα αυτό γιατί συμπίπτει με τη σύσταση της Διερευνητικής Επιτροπής. Είναι σημαντικό η Επιτροπή Μεταφορών να αποφανθεί επί του θέματος και λυπούμε γιατί μόνο γνωμοδότηση μπορούμε να έχουμε και όχι μεγαλύτερη αρμοδιότητα, όπως θα έπρεπε. Συμφωνώ με πάρα πολλά με την κυρία Κάριμα Ντελή και θέλω να επανέλθω στη Διερευνητική Επιτροπή και να πω το εξή. Ενιαία αγορά χωρί εναρμόνιση κανόνων και χωρί έλεγχο, ε, αυτό είναι καταστροφικό για το γενικό συμφέρον. Βέβαια, βολεύει και συμφέρει του κατασκευαστέ, όχι όμω του καταναλωτέ και του πολίτε που υφίστανται την ατμοσφαιρική ρήπανση βλέπουμε για άλλη μια φορά ότι χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη αλλά κυρίως καλύτερη Ευρώπη. Δεν είναι δυνατό ε, την ανάκληση των οχημάτων να την αποφασίζει το εκάστοτε ε, κράτος και όχι το γειτονικό του. Δεν γίνεται ε, να έχουμε γελίες κυρώσεις σε περίπτωση απάτης και τα κράτη-μέλη ουσιαστικά να καταχωρίζουν και να αποκτούν επιστοποίηση για τα οχήματα, ούτε καν εκεί που ε, είναι πιο εύκολο ή που οι κανόνες είναι πιο σαφείς, αλλά στο κράτος μέλος που ασχολείται λιγότερο με αυτούς. Πρέπει να έχουμε τυποποιημένα τεστ που να αποτελούν προσωμείωση των πραγματικών συνθηκών οδήγησης και θα πρέπει να δοθεί ένα τέλος στις ε, ε, στις ε, διάφορες συγκρούσεις συμφερόντων σε όλη αυτή την αλυσίδα πιστοποίησης. Πρέπει ο κάθε φορέας να είναι ανεξάρτητος. Ο έλεγχος και η επιτήρηση και η εποπτεία των αγορών πρέπει να είναι αποτελεσματικός, ανεξάρτητος. Και είναι απολύτως απαραίτητο να διασφαλίσουμε αυτή την ανεξαρτησία. Ακόμα και αν δοθεί πιστοποιητικό, πρέπει το όχημα να παραμένει πληρούν τους όρους και αυτό πρέπει να επιβεβαιώνεται από τους τεχνικούς ελέγχους στη συνέχεια. Έχει αλλάξει χρονοδιάγραμμα και ασκείται πίεση να προχωρήσουμε γρήγορα για την έκθεση αυτή, χωρίς να περιμένουμε τα συμπεράσματα και τα πορίσματα της Διερευνητικής Επιτροπής. Ενώ εμείς θέλουμε να υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο. Δεν θέλουμε να προχωρήσει γρήγορα η γνωμοδότησή μας πριν αποφανθεί η Διερευνητική Επιτροπή. Και χαίρομαι γιατί και οι σκιώδη το ίδιο είπαν είναι σημαντικό να πάμε μέχρι τέλους και να εδραιώσουμε κανόνες που που θα ε, καλύπτουν ό,τι, έχουμε, ό,τι έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα και που θα είναι προς το συμφέρον καταναλωτών και πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σπάχο. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να τονίσω πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό και πόσο ευαίσθητο. Οι συνάδελφοι το έκαναν αυτό άλλωστε. Να πω μόνο το εξή. Ότι να μην επιβάλλουμε, ενδεχομένω. Γιατί υπάρχουν πολλέ ε, υπηρεσίε ε, έγκριση ε, τέτοιων οχημάτων που τηρούν μια χαρά τους κανόνες που είναι επιστοποιημένε, που κάνουν τακτικούς ελέγχους και εποπτεία. Αυτό που λείπει και αυτό που υπάρχει είναι κάποια κενά στην εφιστάμενη νομοθεσία και αυτά θεωρώ ότι θα πρέπει να μας απασχολήσουν όλους ιδιαίτερους για να τα καλύψουμε τα κενά αυτά. Η Καρίνα, Καρίμα προτείνει στην ε, μια τροπολογία περιθμών 14 για τον διαχωρισμό των ε, τεχνικών υπηρεσιών και των ε, υπηρεσιών Έγκριση και των παραγωγών. Πολύ βασικό αυτό. Επίσης θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και το διέγραψε η Καρίμα είναι αυτός ο εκτελεστικός, εκτελεστική νομοθετική πράξη. Έχουμε αρκετή εμπειρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και μετά από αυτά που είπαν και οι συνάδελφοι για την μεγάλη αυτή Ευρωπαϊκή Υπηρεσία που προτείνει και η Καρήμα στην τροπολογία 28. Εδώ θα πρέπει να επιδείξουμε ιδιαίτερη προσοχή, πιστεύω. Ευρωπαϊκή εποπτεία, ναι, με ασφάλεια. Αλλά τώρα να δημιουργήσουμε μια νέα υπερευρωπαϊκή τέτοια υπηρεσία, αυτό με προβληματίζει. Γενικά, θα πρέπει να πω ότι αυτό το peer-to-peer, -peer, όπως όπω οπως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή η αξιολόγηση του ενός κράτους από το άλλο, δεν είναι κάτι το οποίο συνάδει με την εικόνα που έχω για την Ευρώπη. Ποια ρυθμιστική υπηρεσία θα μπορούσε να ελέγξει τη ρυθμιστική υπηρεσία μιας άλλης χώρας. Θεωρώ ότι αυτό θα οδηγούσε σε συγκρούσεις ένα άλλο θέμα. Μίλησε ο κ. για τα ρημουλκούμενα. Υπάρχουν πολλέ μικρομεσαίε επιχειρήσει ε, στην Ευρώπη που παράγουν ε, μικρών σειρών, μικρές σειρές. Θα πρέπει λοιπόν να τα λάβουμε αυτά υπόψη ότι υπάρχουν, ε, υπάρχουν πολλοί μικροί παραγωγοί οι οποίοι και αυτοί θα πρέπει να έχουν μια κάποια ευελιξία και ασφαλώς φυσικά παράλληλα, παράλληλα να ελέγχονται. Αλλά να υπάρχει μία ευελιξία. Μάλιστα, κύριε Μπιμπάου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παίρνω το λόγο για να μοιραστώ μαζί σα ε, δύο ιδέες από τον κύριο Ρικέτ, τον εισηγητή μας, τον Σκιώδη που δεν μπόρεσε να είναι εδώ μαζί μας. Ως ομάδα πολιτική συμφωνούμε να στηρίξουμε τα ευρωπαϊκά πιστοποιητικά και όχι τα εθνικά. Και προτείνουμε να αναβληθεί η εξέταση ε, αυτής της έκθεσης μέχρι ότου βγουν και τα πορίσματα της Ερευνητικής Επιτροπής, να υπάρχει δηλαδή χρονική ε, συμπόρευση των δύο αυτών δράσεων. Η κυρία Αγιάλα Σέντερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ, δεν πρέπει να επιταχύνουμε πριν ολοκληρώσει το έργο της η Ερευνητική Επιτροπή Κοινοβουλευτική για το θέμα αυτό. Και λυπούμε γιατί δεν μπορέσαμε να εμπλέξουμε και την ΙΜΚΟ στο θέμα αυτό. Θα έπρεπε να είχαμε αγωνιστεί για να έχουμε τουλάχιστον κοινή συμμετοχή για τις προτάσεις της κυρίας Ντελή. Δεν είμαστε αφελείς, κανείς δεν είναι αφελείς. Ξέρουμε τι συνεπάγεται για την αυτοκινητοβιομηχανία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Δεν είναι οι Αμερικανοί άγγελοι που έρχονται να μας σώσουν με την περιβαλλοντική τους υπηρεσία. Γερμανοί μηχανικοί είναι αυτοί που ανακάλυψαν αυτή την κατάσταση. Και αναρωτήθηκαν γιατί είναι πιο αποτελεσματικά τα γερμανικά αυτοκίνητα στην Αμερική ως προς αυτό. Οι Γερμανοί μηχανικοί αναρωτήθηκαν και ανακάλυψαν έτσι την απάτη απάτη συγκεκριμένων αυτοκινητοβιομηχανιών, ενδεχομένως γερμανικών, δεν θα πρέπει όλες τι αυτοκινητοβιομηχανίε να τις κατηγορήσουμε σύσσωμε. Στο όταν έχει παλήρια, κάποιοι άλλοι κερδίζουν και ψαρεύουν, κάποιοι άλλοι όχι. Σε κάποιες χώρες συναρμολογούμε μικρά αυτοκίνητα με μικρότερη κατανάλωση και μικρότερο αντίκτυπο. Επομένως, αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Όντως πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές και καλό θα ήταν να μειωθεί η κατανάλωση σε μια πρώτη φάση. Αλλά ούτως ή άλλως έχουμε μικρότερα και πιο ελαφριά οχήματα και άρα έχουμε μειωμένη κατανάλωση. έχουμε ένα θύλακα ευκαιριών, μια ε, μικρή μερίδα αγοράς. Δεν γίνεται οι μικρές εταιρείες να ε, είναι εθνισυγενείς για το αμάρτημα των μεγάλων μητρικών ε, επιχειρήσεών τους. Πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές λύσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε και το Τέσλα. και τελικά είμαστε ανταγωνιστικοί. Και είναι ένας αγώνας, ε, μια μάχη ανταγωνισμού. Υπάρχουν και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Όμως δεν είναι τόσο πράσινα και τόσο θαυμάσια όσο νομίζουμε. Όλα αυτά έχουν σχέση και με τις εθνικές αποφάσεις. Εξού και στις ευρωπαϊκές αποφάσεις στηρίζω αυτό που είπε ο συνάδελφος. Θα είναι πολύ δύσκολο να έχουμε μια κοινή ευρωπαϊκή αρχή Μπορεί αυτό να ευνοήσει τους πολίτες, τους καταναλωτές, να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Απ' την άλλη υπάρχει το ε, βιομηχανικό απόρριτο και η δυνατότητα καινοτομίας και πρέπει να τα προστατεύσουμε όλα αυτά. Υπάρχουν θέματα που είναι εθνικά, εθνικές στρατηγικές αποφάσεις. Το γνωρίζουμε και κανείς δεν είναι αφελής. Λύσεις. Τώρα, να έχουμε την προοδευτικότητα. Δηλαδή να μειώσουμε την κατανάλωση και να μειώσουμε τον αντίκτυπο των εκπομπών, αυτό να γίνει σε μια πρώτη φάση και έχουμε προχωρήσει ιδιαίτερως, έχουμε μειώσει τον αντίκτυπο των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, να μειώσουμε λοιπόν την κατανάλωση και τις εκπομπές, αλλά να μην σφαγιάσουμε την αυτοκινητοβιομηχανία. σε πρώτη φάση δηλαδή να πρημοδοτήσουμε τα μικρά ελαφριά αυτοκίνητα σε μεσοπρόθεσμη βάση. Να υιοθετήσουμε άλλης φύσης μέτρα και σε μακροπρόθεσμη βάση να κάνουμε αυτή τη τεράστια διαρθρωτική και δομική αλλαγή και βοηθώντας πάντοτε τους φορείς. Δεν μπορούμε να ε, κλείσουμε μία αγορά μέσα σε μια νύχτα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κ. Κόχα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόταση τη σε σχέση με το θέμα αυτό. Και ιδιαίτερω επειδή δεν συνεπάγεται επιπλέον κόστος για τον καταναλωτή και την κυρία Ντελή θα ήθελα να ευχαριστήσω. Ωστόσο, κάποια στιγμή με απασχολούν και είμαι αρκετά επικριτικό. Όπω αυτή η ιδέα για μια νέα Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή. Αυτό το είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Επίση, ε, η εισηγήτρια αναφέρεται συχνά στην ε, Volkswagen. Θα ήθελα να σταματήσει κάπως αυτό, όχι ως ε, Γερμανός και μόνο, αλλά επειδή υπάρχουν πολλοί πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες οι οποίες έκαναν παράνομε, πα, παρόμοιες ενωθείς, ίσως και χειρότερες. Ε, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι η αναφορά για, την αυστηρή, για τον αυστηρό διαχωρισμό των παραγωγών, των ελεκτών και των ε, υπηρεσιών αδειοδότησης. Αν θέλουμε να υπάρχει ανεξαρτησία, ασφαλώς και είναι απαραίτητο να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Τώρα, κατά είναι η πρόταση για την ε, ε, ενιαία επιβολή τελών ε, εξυπηρετεί το σκοπό του αυτή διαχωρισμού αυτού, δεν είμαι σίγουρος να σας πω την αλήθεια. Πιστεύω ότι ενδεχομένω να είναι και αντιπαραγωγικός αυτός ο διαχωρισμός. Και αυτός ο περιορισμός στα πέντε έτη που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύω ότι είναι υπερβολικός. Είναι υπερβολικά μικρή αυτή η χρονική περίοδος και προς την κατεύθυνση αυτή θα καταθέσω τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος ε, Ισμαήλ Ερτούκ. Ευχαριστώ πολύ. Και καταρχάς, να σας πω τι λέει η κυρία Γκραπίνη που είναι η συγγητριά μας, γιατί μας ξεχάσατε. Ξεχάσατε το σοσιαλιστή, τη σοσιαλιστρία Σκιώδη. Όχι, κοιτάξτε, νόμιζα το θα έλεγε η κυρία Ριβόλ. Αλλά όχι, όχι, πείτε μας. Και μετά θα παρουσιάσω και τις δικές μου ιδέες για το θέμα αυτό. Come on, speak, boss. Concentration please. Yes, I, I would like to follow, uh, the, the, uh, present now the statement of... Λοιπόν, η δήλωση της κυρίας Γραπίνη. Η δημιουργία ε, μια ευρωπαϊκή τέτοια αρχή για την έγκριση και την εποπτεία τη αγορά ε, είναι καλή ιδέα, αλλά θα προαπαιτούσε χρηματοδότηση σε ένα ξεχωριστό κανονισμό. Υποστηρίζω την αρχή, αλλά δεν πιστεύω ότι μια τέτοια αρχή μπορεί να δημιουργηθεί με τον παρόν κανονισμό. Και εκ παραλλήλου δεν μπορώ να υποστηρίξω την ιδέα μια τέτοια ε, υπηρεσία που θα έχει την αρμοδιότητα για την έγκριση των πράξεων κατεξουδότησης, γιατί σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης, μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει πράξεις εξουσιοδότησης και πιστεύω ότι το Ελεκτικό Συνεδρίο ή οποιοδήποτε ειδικό σώμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έπρεπε να κάνει τέτοιου έλεγχου για τα κρατημέλη μέχρι ότου δημιουργηθεί μια τέτοια Ευρωπαϊκή Αρχή. Ο έλεγχο θα πρέπει να έχει στο στόχαστρο και τι αρχέ των κρατών μελών και να καθορίζει κατά πόσον συνάδουν με τον νόμο η έλεγχη, αλλά και τα κρατημέλη για να διαπιστώνεται κατά πόσον εφαρμόζονται σωστά η νομοθεσία. Και πιστεύω ότι χρειάζεται ε, καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διάφορων κρατών μελών και των σχετικών υπηρεσιών για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων. Επίσης, ε, γίνονται έρευνες ε, από τους επιστήμονες για να καταλήξουμε σε στοιχεία βάσει των οποίων θα μπορέσουμε να κάνουμε τι νομοθετικέ προτάσει. και αυτό θα πρέπει να γίνει παράλληλα με τι έρευνε που γίνονται από τι αρχέ έγκρισης τύπου από τη, τα κράτη-μέλη. Θα συζητήσουμε λοιπόν τα θέματα αυτά και με τα μέλη τη ομάδα μου για να δούμε πώ θα μπορέσουμε να έχουμε και τη σωστή προστασία αλλά και να μην επιβαρύνουμε τι μικρέ επιχειρήσει. Αυτά λοιπόν λέει η συνάδελφο Γκραπίνη. Τώρα, εγώ να πω και εγώ προσωπικά δύο λόγια γιατί είμαι ένα από τα μέλη της Ερευνητικής Επιτροπής και πιστεύω ότι τα πιο σημαντικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Ερευνητική Επιτροπή και γενικώ δηλαδή, είναι τρία στοιχεία. Καταρχάς, έλεγχος διαφάνεια. Και ο εκ των υστέρων έλεγχος. Και τώρα θα μιλήσω και γερμανικά γιατί είναι λίγο πιο απλό να τα πω τα τεχνικά αυτά ζητήματα στη μητρική μου γλώσσα. Σε ό,τι αφορά την ε, η ποιότητα των υπηρεσιών αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να υπάρχει ένα πιο νέο επίπεδο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και η ιδέα για μια ευρωπαϊκή υπηρεσία είναι καλή και ευκταία, αλλά θα πρέπει να συμμετέχουν στην διαμόρφωση των υπηρεσιών αυτών και τα κράτη-μέλη. Και αυτά θα πρέπει να είναι δημόσια προσβάσιμα προκειμένου να είναι γνωστές και οι ατασταλίες και τα προβλήματα που παρουσιάζονται. Και αυτό αποτελεί και μία προϋπόθεση και αυτό που θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό είναι να έχουν πρόσβαση σε αυτά και ανεξάρτητες τρίτες αρχές. Θα πρέπει λοιπόν να διορθωθεί η σημερινή κατάσταση. Η γενικότερη κατεύθυνση του να περάσουμε από μια οδηγία σε κανονισμό είναι σωστή για να για να μην έχουμε 28 διαφορετικά συστήματα και 28 διαφορετικές μορφές τέτοιων προτύπων ποιότητας. Αυτό δεν είναι πλέον βιώσιμο. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε. Και μας επηρέασε και το πρόσφατο σκάνδαλο με τις εκπομπές. Γι' αυτό λοιπόν πολλά ακόμα έχουμε να κάνουμε. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος, μπήκα και εγώ στην ημερήσια διάταξη να πω δύο λόγια η κυρία Γελασάντερ μίλησε για διακύβευση για τον της απασχόληση. Μα ποιο τη υπονόμευσε τι θέσει απασχόληση, οι αυτοκινητοβιομηχανίε. Αυτέ έπεσαν εν κινδύνο τι θέσει απασχόληση αυτέ. Αυτέ εξαπάτησαν τον κόσμο και έβαλαν σε κίνδυνο τελικά τη ζωή του κόσμου και από αυτού, κανείς δεν έχει προσαχθεί ακόμα, κανείς δεν έχει κρυθεί ενοχώ. Ως τώρα ακόμα τίποτα δεν έχει γίνει, μόνο συζητιούνται όλα αυτά. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι υποπροστασία, γιατί φυσικά πρόκειται για συνεργασία μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών και των πολιτικών ηγεσιών. Και αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είναι μόνο η Volkswagen, έχει απόλυτα δίκιο ο Dieter Koch όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες κάνανε τέτοιες απάτες και ήταν οι Γερμανοί, οι μηχανικοί το που υπογράμμισαν αυτό. Αλλά δεν ε, πήγαν στι ΣΥΠΑ για να υποδείξουν ότι γινόντουσαν οι απάτες αυτές. Όχι, στην αρχή το επέδειξαν και το κατέδειξαν αυτό προς την ε, γερμανική κυβέρνηση, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό πριν από 5-6 χρόνια και δεν έγινε τίποτα, καμία δεν ήταν η αντίδραση. Ε, λοιπόν, κάποιες συνέπειες θα πρέπει να υπάρξουν από την Volkswagen με 300 ευρώ ανά αυτοκίνητο θα μπορούσαν να πληρούν τα πρότυπα και τις οριακές τιμές. Ε, μα για 300 ευρώ δηλαδή ένα αυτοκίνητο τελικά τώρα ε, πληρώνουν ε, και θα πληρώσουν πρόστιμα ύψους δισεκατομμυρίων. Ούτε οικονομικά δεν βγάζει νόημα αυτό. Και από ό,τι φαίνεται όλοι το ήξεραν, γιατί όταν εξάσπασε το πρώτο σκάνδαλο όλοι σιώπησαν. Γιατί κανονικά, ξέρετε, ε, αν ε, ήταν ε, αθώοι όλοι οι υπόλοιποι, θα είχαν βγει και θα μένονταν και θα τους κατηγορούσαν και θα λέγανε ότι κοιτάξτε εμείς που τηρήσαμε τα πρότυπα κτλ. κτλ. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία. Ούτε οι Ιταλοί, ούτε οι Γερμανοί, ούτε οι Ισπανοί, κανείς δεν τηρήσει τα πρότυπα αυτά. Όλοι εξαπάτησαν. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές. Ε, κοιτάξτε, τώρα δεν λέω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια τεράστια ευρωπαϊκή αρχή, αλλά θα πρέπει να έχουν τις ε, αρμοδιότητα να κάνουν δειγματολεπτικούς ελέγχους για να διαπιστώνουν κατά πόσον στέκουν τα στοιχεία τα οποία υποβάλλονται και αν υπάρχουν ε, προβλήματα, αν υπάρχουν αν να τι επισημαίνουν. Αυτό φυσικά είναι κρατική κρατικό καθήκον. Μιλήσαμε πάρα πολύ και για θέματα ανεξαρτησίας. Όλοι είμαστε υπέρ ασφαλώς. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει και οικονομική, χρηματική ανεξαρτησία. Γιατί είδαμε στην Ευρώπη κάποιοι τύποι αυτοκινήτων πήγαν προς το Λουξεμβούργο, προς τη Γερμανία, προς την Γαλλία. Άνω ίδρυμα δηλαδή, Άνω υπηρεσία. Είμαι τόσο ανεξάρτητος που έρχεται προς εμένα η αυτοκινητοβιομηχανία. Ε, δεν θα είμαι αυστηρός γιατί ξέρω ότι εξαρτάται και η επιβίωσή μου από την εκάστοτε εταιρεία. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται απόλυτη ανεξαρτησία. Στη Γερμανία να σας πω ότι αν είχαμε επενδύσει στη Γερμανία ένα ευρώ στην ε, υπηρεσία αυτή θα μπορούσαμε να έχουμε μια πραγματική ανεξαρτησία. Όχι, θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει η οικονομική ανεξαρτησία, όπως και η στη Γερμανία, η, το αντίστοιχο κτέο, που είναι απόλυτα ανεξάρτητο ως υπηρεσία. Αυτό θα πρέπει να συμβεί. Άρα, θεσμική ανεξαρτησία, αλλά βασικά και κυρίως και οικονομική ανεξαρτησία. Ιδάλλως θα επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα και νομίζω ότι κανείς δεν το επιθυμεί αυτό. Κάποιοι θα είχαν ίσως το όνειρο να το κάνουν αυτό, να κάνουν δηλαδή μια απάτη και να μην τους πιάσουν, αλλά εμείς τι θέλουμε. Και το βλέπω τώρα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή είναι η για το ε, σχέδιο έκθεση. πρόκειται για τροπολογίε και αλλαγές ε, που συμβαδίζουν με τα όσα έχει προτείνει στο σχέδιο της Κομισιόν. Ο στόχο μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι το σύστημα έγκριση τύπου θα είναι πιο στεναρό και αποδοτικό αποτελεσματικά και πιο αξιόπιστο στην Ευρώπη. Πιστεύουμε ότι το κείμενο της έκθεσης ε, ανταποκρίνεται σε αυτές τις προσδοκίες και γι' αυτό και είμαστε ευχαριστημένοι που βλέπουμε το σχέδιο το το, της τροπολογίας. Επίσης είναι εξίσου σημαντικό η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο με τις, Επιτροπές σας να στέλνουμε το ίδιο ισχυρό και ξεκάθαρο μήνυμα ότι χρειάζονται θεμελιώδεις αλλαγές στο σύστημα και αυτό κάνει και η έκθεσή σας ότι δηλαδή δεν μιλάμε μόνο για καλοπιστικές ε, ε, αλλαγές αλλά για ε, εκβάθρων ε, αλλαγή. Το καλωσορίζουμε αυτό. Δεν θα συζητήσουμε τώρα σήμερα τις λεπτομέρειες των τροπολογιών. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε κάποιες προτάσεις, σε κάποιες αλλαγές ε, αυτό που εμείς μπορούμε να εγκρίνουμε είναι όλες οι τροπολογίες που κατευθύνονται προς την μεγαλύτερη διαφάνεια, την καλύτερο διαχωρισμό των ρόλων των φορέων στη διαδικασία έγκρισης τύπου. Επίσης κατανοούμε την περιβαλλοντική ευαισθησία που αντικατοπτρίζεται σε διάφορες τροπολογίες και είμαστε της άποψης πως αυτός είναι ο σωστός τρόπος να τονίσουμε τη σημασία των περιβαλλοντικών θεμάτων και τέλος ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς και των διαδικασιών επιβολής είναι κάτι με το οποίο συμφωνούμε. Χωρίς να μπω λοιπόν σε λεπτομέρειες πιστεύουμε ε, ότι είναι πρόσδεκτες οι τροπολογίες αυτές και Είμαστε στη διάθεσή σας για να δωσουμε διευκρινησει διευκρινήσεις. Υπάρχουν ωστόσο δύο-τρία σημεία που θα ήθελα να τονίσω, όπου η Κομισιόν έχει κάποιες ανησυχίες. Το πρώτο αφορά την δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής. Αυτό που προτείναμε είναι το σύστημα της εποπτείας και της ε, ανεξάρτητης εποπτείας που πιστεύουμε αρκεί ώστε να εξασφαλίσουμε πως ε, γίνεται όντως η εποπτεία της αγοράς από τα κράτη-μέλη. Συμφωνούμε επίσης και με την αρχή της ανεξαρτησίας, όπως την υπογραμμίζει η συγγήτρια, αλλά η ανεξαρτησία είναι μία από τις προϋποθέσεις. Υπάρχει και το θέμα του προϋπολογισμού, της τελέχωσης του χρόνου. Ε, πιστεύουμε λοιπόν πως η ανεξαρτησία θα πρέπει να ενταχθεί περισσότερο στο σύστημα, αλλά όχι απαραίτητο μέσω της δημιουργίας ενός ανεξάρτητου θεσμού. Ο μας, δεύτερος μας αφορά τον χρονισμό της πρότασης. Αναγνωρίζουμε και εκτιμούμε την εργασία της Επιτροπής ΕΜΙΣ και τα πορίσματα της, αλλά θέλω να μιλήσω για το πόσο επίγουσα είναι η μεταρρύθμιση αυτού του συστήματος που δεν αποδίδει, ε, δεν λειτουργεί επαρκώς και που δεν είναι επαρκώς ευαίσθητος απέναντι στην προστασία του καταναλωτή, οπότε οποιασδήποτε προστασία δεν είναι προς όφελος. Και δεν μιλάμε ούτε να βιαστούμε, ούτε να ε, γίνει εις βάρος της ποιότητας, αλλά σίγουρα θα πρέπει να επεξεργαστούμε αυτή την πρόταση όσο γίνεται πιο σύντομα. Τελευταίο σχόλιο αφορά τους κανόνες για τις εκπομπές. Πιστεύουμε πως οι αλλαγές είναι δίκαιες, αλλά η νομοθεσία έγκρισης τύπου δεν είναι το κατάλληλο σημείο για να αντιμετωπίσουμε άμεσα τα θέματα του μηχανισμού αλλίωσης ή της στρατηγικής προστασίας των κινητήρων. Αυτά ήδη αναφέρονται στις οδηγίες που αφορούν τα θέματα εκπομπών ε, και πάλι λοιπόν είμαστε στην διάθεσή σας για να βρούμε τις καλύτερες διατυπώσεις και προτάσεις. Αλλά εν γέννη στηρίζουμε την έκθεση που έχει σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει πάλι γητρία. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι διότι η Επιτροπή λέει σήμερα ότι πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα ενώ η παθητικότητά της είναι εμφανέστατη 10 χρόνια για το φάκελο αυτό, για την υπόθεση αυτή, κάτι το οποίο είναι αρκετά σοβαρό. Εγώ λοιπόν λέω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό το ζήτημα αυτό και πρέπει να πάρουμε το χρόνο που χρειάζεται για να μην χρειαστεί να ξανααναθεωρήσουμε την νομοθεσία και μέσα σε ένα-δύο χρόνια να ξαναανακαλύψουμε τα μου σκάνδαλα. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται τέτοια πράγματα. Θέλουμε να συνεργαστούμε στενά με την ΙΜΚΟ και την ΕΝΒΗ, τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές για την Προστασία του Καταναλωτή, την Εσωτερική Αγορά και των Περιβάλλων. Αποκαλύφθηκε αυτό το σκάνδαλο και αν η έλεγχη δεν είναι πραγματική, αποτελεσματική και αποδείχθηκε ότι είναι αναποτελεσματική για το ε, μονοξίδιο του αζότου Αν δεν μπορούμε να κάνουμε σωστούς ελέγχους για το μονοξίδιο του αζότου, τότε ούτε σε θέση θα είμαστε να κάνουμε σωστούς ελέγχους για την ασφάλεια ή την οδική κυκλοφορία. Είναι υγειονομικό το σκάνδαλο μεταξύ άλλων. Από εκεί και πέρα. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό για τον έλεγχο και την ανεξαρτησία. δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους, ε, στους εαυτούς μας να μην υπάρχουν έλεγχοι. Εγώ προτείνω την μεγάλη αυτή ευρωπαϊκή υπηρεσία. Άκουσα την ε, Επίτροπο Φερχάγγελ και έχω ερωτηματικά. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι πραγματικά ανεξάρτητη σήμερα. Με προβληματίζει αυτό. Έχετε δίκιο τα βασικά ζητήματα θα πρέπει να ε, θίγονται σε αυτή την έκθεση. Ποιος αποφασίζει. Πώς γίνεται η επαλήθευση. Σε κάθε περίπτωση και συμπεραίνω και ολοκληρώνω με αυτή την παρατήρηση θεωρώ ότι δεν μπορεί να γίνεται πλέον δεκτό το επιχείρημα της ανεργίας των μισθωτών, των εργαζομένων, αν ασχοληθούμε με την αυτοκινητοβιομηχανία. Δεν γίνεται να μην ασχολούμαστε με την αυτοκινητοβιομηχανία επειδή θα μπορεί να κινδυνεύσουν κάποιοι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι θύματα του σκανδάλου της αυτοκινητοβιομηχανίας, γιατί τους στείνουμε στο τοίχο με ε, απατηλά λογισμικά που εξαπατούν, ενώ δεν φταίνει οι εργαζόμενοι και πρέπει να τους μετατρέψουμε, να τους τρέψουμε ε, προς τις ενέργειες του, ε, του αύριο, δηλαδή να μπορούν να φτιάχνουν αυτοκίνητα με υδρογόνο, με άλλες πηγές ενέργειας πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Οι εργαζόμενοι που θα είναι τα πρώτα θύματα, γιατί με παθητικό τρόπο παρατηρούμε όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Σίγουρα θα είναι οι συζητήσεις ε, τεταμένες. Το θέμα γύρει πολλά πάθη. Όμως, δυστυχώς δεν αφορά μόνο τη Volkswagen, αλλά πάρα πολλούς κατασκευαστές. Ο σκοπός είναι να μην έχουμε πλέον diesel gate στην Ευρώπη και να δείξουμε εμείς οι νόμοθέτες ότι είμαστε σε θέση να θεσπίσουμε κανόνες που μπορούν να τηρούνται πρώτον και δεύτερον ότι ξαναφέρνουμε στο προσκήνιο τα δικαιώματα των καταναλωτών οι οποίοι ουσιαστικά τους έγδαραν οι αυτοκινητοβιομηχανίες, τους κατάκλεψαν και πρέπει να συντάξουμε μια νέα ιστορία της Ευρώπης, να μπορούμε να δείξουμε ότι η Ευρώπη βρίσκεται για να προστατεύει τους πολίτες, ε, ειδικότερα στο πεδίο της ε, ατμοσφαιρικής ρήπανσης και της μόλυσης του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Προθεσμία για τις τροπολογίες 13 Σεπτεμβρίου, το η το μεσημέρι. Και έτσι λοιπόν κανονικά θα είχαμε ολοκληρώσει την συνεδρίασή μας και συνεχίζουμε κλεισμένο των θυρών με τους συντονιστές.